Good morning, ladies and gentlemen, again. Now we are together, all of us. Καλημέρα και κύριοι και πάλι. Είμαστε λοιπόν όλοι μαζί εδώ για τη συμμετοχή σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική αλλά και ευχάριστη συνεδρίαση. Οποιαδήποτε συνεδρίαση με του μέλη του Επιτροπή είναι ευχάριστη. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να ευχαριστήσουμε για του συναδέλφου από την Επιτροπή Ρέτζι και εκτιμούμε ιδιαίτερα την ευκαιρία να συζητήσουμε την 7η έκθεση για τη συνοχή από κοινού με του συναδέλφου από την Επιτροπή των Περιφερειών. Να καλώ ορίσω και τον κύριο Όσβαλτ, να τον συγχαρώ για την εκλογή του ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, ΚΟΤΕΡ Ελπίζω να συνεχίσουμε την επικοινωνική συνεργασία. Να καλωσορίσω και την Επιτροπό Κρέτσου. Με χαρά σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Ήταν δύσκολο να φτάσετε στο Κοινοβούλιο από ό,τι καταλάβαμε. Για όλους μας βέβαια. Η πρόσβαση ήταν δύσκολη για όλους μας σήμερα το πρωί. Με χαρά όμως θα ακούσουμε τα όσα έχετε να μας πείτε και θα ακούσουμε τις πληροφορίες για την 7η έκθεση για τη συνοχή τις απόψεις σας, ε, τα μηνύματα τα οποία έχετε να διαβιβάσετε προς την Επιτροπή των Περιφερειών και προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην αρχή της συνεδρίασης ε, υποσχέθηκα ότι θα είμαι πάρα πολύ σύντομη στην εισαγωγή μου γιατί πιστεύω πιο σημαντικό είναι να ακούσουμε την Επιτροπό. Να πω μόνο το εξής στην Επιτροπή Ρέτζη είμαστε πάρα πολύ επικεντρωμένοι, πολύ φιλόδοξοι και ιδιαίτερα κινητοποιημένοι σε ό,τι αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής ως πολιτική πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις πτυχές της μελλοντικής πολιτικής συνοχής δημιουργώντας και παράγοντας εκθέσεις εφαρμογής ε, και υλοποίησης. Ήδη δημοσιεύσαμε το όραμα για το μέλλον της πολιτικής συνοχής με την ε, ε, έκθεση πρωτοβουλίας μας Building Blocks για την πολιτική της συνοχής ακρογωνία ηλίθεια αν θέλετε της ευρωμελευτικής πολιτικής για τη συνοχή και σε όλες τις συναντήσεις μας και συνεδριάσεις μας συζητήσαμε τα πολύ σημαντικά τα θέματα τα οποία άπτονται της πολιτικής συνοχής συμφωνήσαμε και σε ό,τι αφορά κάποια βασικά μηνύματα για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πολιτική συνοχή καταρχάς, χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες του παρελθόντος για τον καλό σχεδιασμό της μελλοντική πολιτικής συνοχής που προσανατολίζεται στις ανάγκες του Ευρωπαίου πολίτη. Το αναφέραμε αυτό και χθες κατά την ανακτήρια συναντρίαση. Οι ανάγκες του πολίτη θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο κάθε προσπάθειά μας. Και θα πρέπει όλες οι αλλαγές και όλες οι βελτιώσει τη πολιτική συνοχή να προσαρμοστούν ακριβώς στις ανάγκες του Ευρωπαίου πολίτη. Κατά δεύτερον, πιστεύουμε πραγματικά ότι υπάρχουν πολύ πιο πολλές ευκαιρίες σε ό,τι αφορά τον συντονισμό και τη στενότερη συνεργασία μεταξύ πολιτική συνοχή και των άλλων πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καλό μείγμα λοιπόν μεταξύ πολιτική συνοχή και πολιτικών στην εκπαίδευση, καινοτομία, κοινωνικέ πολιτικέ, εμπόριο, ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένη προφανώ και τη πεθύρικη ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι στο μέλλον βιώσιμη, ευέλικτη η πολιτική συνοχής επικεντρωμένη στις ανάγκες του πολίτη και στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει καινούργιε προκλήσεις. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτική συνοχής να προσαρμοστεί στις τρέχουσες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μεταναστευτική κρίση, φυσικές καταστροφές, κλιματικά ζητήματα, οικονομικά προβλήματα ζητήματα ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, η υψηλά ποσοστά ανεργία σε πολλές περιφέρειες, όλα αυτά αποτελούν προκλήσεις και η πολιτική συνοχής έχει ενδογενώς την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές. Αυτή είναι η τοποθέτησή μας. Και με μεγάλο ενδιαφέρον, συμπληρωματικά προς την δική μας δουλειά, θα ακούσουμε την άποψη της επιτροπή των Περιφερειών και την άποψη φυσικά της Επιτρόπου για την 7η εκθέση για τη συνοχή. Βάζω τελεία στο σημείο αυτό, σα το υποσχέθηκα. Ξέρετε ότι μπορεί να μιλήσω, μπορώ να μιλήσω πολύ παραπάνω, αλλά θα δώσω το λόγο στον κύριο Οσβάν καταρχά για να συνεχίσει τα εισαγωγικά σχόλια. Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Έχω την ομιλία μου εδώ μπροστά, αλλά είστε τυχεροί δεν έχω μαζί τα γυαλιά μου. Δεν έχουμε και χρόνο. Νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα με τις δηλώσεις της κυρίας Μιχαήλοβα. Ευχαριστώ όλους τους παρευρισκόμενους συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής για το πολύ σημαντικό αυτό έγγραφο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Μιχαήλοβα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, κύριο Κατάνο από την Πρόεδρια της Επιτροπής Κότερ θα συνεχίσουμε το έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη εδώ και πιστεύω ότι ήταν καλή απόφαση να συναντηθούμε σε ειδικέ περιστάσεις όπως η σημερινή. Ο κανονισμός ε, κανονικά από ό,τι ξέρω θα ολοκληρωθεί σε 8 μήνες. Έχουμε πολλά ζητήματα λοιπόν να εξετάσουμε ακόμα. Τον κύριο Σπυρίδων του πρώτο αντιπρόεδρο θα ήθελα να σας αισθήσω. Και βάζω και εγώ τελεία στο σημείο αυτό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Χάσαμε χρόνο σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Το λόγο λοιπόν τώρα έχει η Επιτροπή Κρέτσο. Σα καλωσορίζουμε. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη Πρόεδρε τη Επιτροπή Ρέτζη και τη Επιτροπή Κοτέρ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή Κοτέρ, καλημέρα σα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση να παρευρεθώ σε αυτή την παραδοσιακή κοινή συνεδρίαση μεταξύ Ρετζή και Κοτέρ ε, των ε, περιφερειών και των πόλεων ουσιαστικά. Ξέρετε ότι εχθές είχαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο το οποίο δημοσιεύθηκε την 7η έκθεση συνοχής που ε, προκύπτει από την απέτηση να αναφέρουμε πώς έχει εξελιχθεί η πολιτική συνοχής ε, στο πρόσφατο παρελθόν και βεβαίως υπάρχει και πολύ τροφή διασκέψη η οποία έχει προκύψει από αυτή την έκθεση. Όπως είπε ήδη λοιπόν η πρόεδρος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε το θέμα αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι ποτέ, διότι μπαίνουμε στην τελευταία φάση στην προετοιμασία του μέλλοντος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ξέρετε ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε ήδη ότι το πρώτο σχέδιο του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο το Μάιο. Επομένως έχουμε περίπου 8 μήνες για διαπραγματεύσεις ξεκινήσαμε τη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή των ε, Περιφερειών και νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να δούμε τι πρέπει να γίνει και μόνο ε, κατόπιν αυτού να δούμε πώς θα πρέπει να γίνει και τι κονδύλια απαιτούνται. Κατά την άποψή μας αυτό το οποίο απαιτείται Δεδομένου ότι έχουμε και λόγους να είμαστε αισιόδοξοι, διότι υπάρχει και πάλι ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία και δημιουργούνται θέσεις εργασίας, Αλλά υπάρχουν και φόβοι οι οποίοι προέκυψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ε, της παγκοσμιοποίησης και της κλιματικής αλλαγής όλα αυτά δεν έχουν εξαφανιστεί και αντανακλώνται στη ζωή των ανθρώπων και στα εκλογικά αποτελέσματα ε, σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει ε, μυσαλλοδοξία και εσωστρέφεια και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μάχη από κοινού προκειμένου να περιορίσουμε αυτή την ελληνεγκή που ε, ε, να αναπτύξουμε μάλλον την αλληλεγγύη που είναι αυτή η οποία ε, συνδέει την Ευρώπη. Η έβδομη έκθεση για την πολιτική συνοχή μας δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού πληθυσμού που θεωρεί ότι παραγωνίζεται παρά τις δυνατότητες ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τα τελευταία 10 χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να αντιληφθούμε ότι δεν είναι τα πράγματα ίδια για όλους. Εξακολουθούν να υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες έχουν χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι είχαν πριν από την κρίση και βεβαίως πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν διαιρέσεις και φόβοι στην κοινωνία μας και να βρούμε έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη λοιπόν την ε, περιφερειακή και τοπική διάσταση, διότι σε πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες οι άνθρωποι είναι φτωχότεροι από ό,τι ήταν πριν από την κρίση, όπως σας είπα. Δυστυχώς, σε πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες ε, ο κόσμος δεν έχει άλλη επιλογή, δεν μπορεί να βρει μια αξιοπρεπή θέση εργασίας, πρέπει να εγκαταλείψουν τις οικίες τους διότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες στην περιφέρειά τους. Και αυτό φυσικά είναι το πιο σημαντικό στις λεγόμενες μεταβατικές περιφέρειες σε περιοχές οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την βιομηχανική μετάβαση. Από την Ανατολή λοιπόν προς τη Δύση, από τις περιοχές της Υπέθρου σε διάφορες περιφέρειες και πόλεις, ο κόσμος ε, αντιμετωπίζει προβλήματα και υπάρχουν ε, στάσιμοι μισθοί, υψηλή ανεργία ε, και καθόλου παραγωγικότητα. Κατά την άποψή μας, περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε μάχη για να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες και να βεβαιωθούμε ότι κάθε Ευρωπαίος έχει πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες όπου κι αν διαμένει. Γι' αυτό και Είμαι πεπισμένη περισσότερο από ποτέ ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τη σύγκληση, τη χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ και πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και τις ίσες ευκαιρίες σε όλες τις περιφέρειες. Κατά την άποψή μου χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και τη χρειαζόμαστε παντού. Τώρα, προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί η πολιτική συνοχή όταν η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει νέε προτεραιότητες και δεδομένου ότι επικρίνεται και η πολιτική μας ε, διότι είχε μια βραδία αρχική πορεία. Αυτή είναι μια αλήθεια την οποία πρέπει να παραδεχθούμε και νομίζω ότι τα πάντα θα πρέπει ε, να ληφθούν υπόψη και να κάνουμε ό,τι μπορούμε τους επόμενους μήνες ε, και να αμφισβητήσουμε το ρόλο των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών ε, για την δέσμευσή τους για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, διότι όπως ξέρετε εμείς είμαστε εδώ για να ε, εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση και τη διαμεσολάβηση, αλλά η εφαρμογή είναι 100% ευθύνη των κρατών μελών. Και εδώ δυστυχώς ε, τα στοιχεία δεν είναι πάρα πολύ καλά για το συγκεκριμένο δημοσιονομικό πρόγραμμα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής ε, πολιτική την οποία πολλές φορές αντιλαμβάνεται λάθος ο κόσμος και ε, παρά τις επικρίσεις ε, φαίνεται να λειτουργεί. Και λειτουργεί διότι δημιουργεί σύγκληση όταν τα οικονομικά μέσα επιτρέπουν να έχουμε τα μακροοικονομικά ε, αποτελέσματα που επιθυμούμε. Λειτουργεί διότι... Ε, τηρεί την υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες ε, πόσιμο νερό, ευρυζωνικά δίκτυα, οδικά δίκτυα, αξιοπρεπείς ε, μεταφορές και συγκοινωνίες, ε, σχολεία, νηπιαγωγία, νοσοκομεία, διότι αντλεί γνώσει από το τοπικό επίπεδο και τι προσαρμόζει ε, σε έργα τα οποία ελοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Συνεργαζόμαστε για να έχουμε συνεργασία δημόσιου τομέα επιχειρήσεων και κοινωνία των πολιτών και κατά την άποψή μου η πολιτική αυτή είναι η πιο προβεβλημένη και είναι αυτή η οποία ε, δίνει απτά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Βεβαίως δεν είμαστε τέλειοι και υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Ε, το έχουμε συζητήσει αυτό και το ε, ε, συζητούμε εδώ και μήνες, αποτελεί στοιχείο προβληματισμού και προσπαθούμε να βρούμε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες για την μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής. Ο κοινό στόχος είναι η μεταρρύθμιση να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους δικαιούχους, δηλαδή για τον πληθυσμό υπάρχουν τέσσερις βασικοί πυλώνες για την πολιτική συνοχή του μέλλοντος κατ' εμέ. Ο πρώτος πυλώνας ε, είναι η εμπιστοσύνη και έγινε χθες ε, η ε, τελετή έναρξης και συζητήσαμε για την εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη μεταξύ θεσμών και πολιτών και ε, φυσικά, όπως είπα, καταμερισμός των ε, ε, βαρών σημαίνει καταμερισμός των ευθυνών, αλλά και καταμερισμός εμπιστοσύνης. Για το διάστημα 2014-2020, ξέρετε ότι καθορίστηκαν κάποιες διαδικασίες για να καθορίσουμε συστήματα ελέγχου και διαχείρισης για να έχουμε και περισσότερη αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τώρα έχουμε την το σύστημα διασφάλισης. Ε, το παρόν σύστημα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να παραμείνει σε εφαρμογή και να αρχίσει να ισχύει από την πρώτη στιγμή. Επίσης, ε, αυτό σημαίνει ότι ε, είναι και συνειδιοκτησία η κάθε πολιτική που εφαρμόζεται και στο σχεδιασμό αλλά και στην εφαρμογή της. Οτιδήποτε έγινε στη διάρκεια της κρίσης δεν αιτιολογείται πλέον. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο εθνικής συγχρηματοδότησης που αντανακλά το ρόλο της κοινή ευθύνη του εθνικού προπολογισμού και η πολιτική συνοχή να εφαρμόζεται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, οι πληρωμές αυτή τη στιγμή βασίζονται στο κόστος των έργων και... Ε, καταβάλλονται ανάλογα με τα τιμολόγια. Θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά αυτό το σύστημα, ε, να έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα βασίζεται στο λογαριασμό, αλλά στο κατά πόσον πληρούνται οι προσυμφωνημένες προϋποθέσεις. Υπάρχουν θέματα όπως η καινοτομία, η ενεργειακή απόδοση, όπου θα μπορεί να είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την απόδοση. Ε, συζητάμε πολύ ε, το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις για το Brexit, ε, δεν ξέρουμε κατά πόσον τα κράτη-μέλη θα είναι διατεθειμένα να συμπληρώσουν το κενό που δημιουργείται, δεν ξέρουμε κατά πόσον θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στα αποτελέσματα και στις επιδόσεις μας. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε επιτύχει πολύ μεγάλη πρόοδο, κυρίως ε, στο πλαίσιο των επιδόσεων ε, και της αιρεσιμότητας ε, και αυτά όλα σχεδιάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτη και κατά την άποψή μου αυτή τη φορά θα πρέπει να πάμε έτη περαιτέρω. Για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να θεζητήσουμε είναι πού θα πρέπει να δαπανηθούν τα κονδύλια. Πιστεύω ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να επικεντρωθεί σε λιγότερους τομείς πολιτικής από ό,τι αυτή τη στιγμή αυτό σημαίνει ότι θα γίνει πιο αποτελεσματική και θα αυξήσει και την προβολή των πολιτικών μας. Ε, Ίσως ε, θα μπορούσαμε να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι πολιτικοί στόχοι, να έχουμε ένα μικρότερο σύνολο στόχων που οδεύουν σε συγκεκριμένους πολιτικές και να έχουμε και τομεακούς στόχους. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ε, και πώς μπορούμε να ε, εντείνουμε την υποστήριξη των διαστροτικών μεταρρυθμίσεων. Οι δημόσιες επενδύσεις είναι πιο σημαντικές όταν υπάρχει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις περί τούτου παρέχουμε θετικά κίνητρα στην πολιτική συνοχής και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσει αυτό. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει και θα πρέπει να το συζητήσουμε δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να είναι εκτός ε, ή υπό την ε, πολιτική συνοχή. Θα πρέπει λοιπόν να συζητηθεί και να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια για το στόχο αυτό. Αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει σχέση μεταξύ πολιτική συνοχή και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ξέρετε ότι αυτό ήταν και στο έγγραφο προβληματισμού για την ε, εμβάθυνση τη οικονομική και νομισματική Ένωση και πολύ ευχαριστώ να ακούσω και τι απόψει για το θέμα αυτό. Τέλος, θεωρούμε ότι θα πρέπει να άρουμε όλους τους μηχανισμούς που συνέβαλαν στην καθυστέρηση της εφαρμογής στη διάρκεια της συγκεκριμένη προγραμματικής περίοδου, ε, να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία, ε, ξεκινώντας από την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση σε δύο χρόνια, αντί για τρία χρόνια που έχουμε τώρα. Διότι διαπιστώνω ότι σε πολλά κράτη-μέλη αυτή η τριετία σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία βιασύνη για να εφαρμοστούν τα προγράμματα και επομένω ε, χάνεται πολύτιμο χρόνος. Ο τρίτος πυλώνα αφορά την ευελιξία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στη διάρκεια αυτής της τριετίας αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές ε, αναπάντεχες ε, προκλήσεις, ε, φυσικές καταστροφές, ο σεισμός στην Ιταλία, η περίπτωση της Βαλονίας της Κατερπίλαρ, ε, και επομένως ε, ξέρετε ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει ξαφνικές πολύ μεγάλες ε, αλλαγές λόγω της παγκοσμιοποίησης ή της της εισρωής προσφύγων. Γνωρίζουμε λοιπόν ε, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένες ε, προτεραιότητες χρηματοδότησης για την ε, επταετία αυτή και πολύ συχνά είναι πολύ δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή και από πολιτική σκοπιά. Μία απλή λύση θα ήταν να έχουμε ένα αποθεματικό για τη συνοχή και όταν προκύπτουν επίγουσες καταστάσεις να χρησιμοποιείται αυτός ο μηχανισμός ταχείας χρηματοδότησης. Έτσι θα είναι πολύ πιο ευέλικτα τα πράγματα και η απαραίτητη ευελιξία θα πρέπει να εξευρεθεί αλλού με τις ε, αντίστοιχες δημοσιονομικές ε, συνέπειες τις οποίες φαντάζεστε. Θεωρώ ότι η ευελιξία θα μπορούσε να ρυθμιστεί με ένα πιο απλό ρυθμιστικό πακέτο και αυτό είναι και ο τέταρτος πυλώνας, η απλοποίηση. Η απλοποίηση ήταν στόχος από την αρχή της θητείας μου. Προσβλέπω και ε, στην έγκριση του κανονισμού Omnibus από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι από τις 4 Ιανουαρίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη νέα δέσμη μέτρων που έχει συμπεριληφθεί στον κανονισμό Omnibus, ε, Omnibus την απλοποίηση των επιλογών κόστους, ε, το συνδυασμό μεταξύ των κονδυλίων του Ταμείου Στρατηγικής Ανάπτυξης και του ΕΣΥΦ ε, και χρήση κονδυλίων για τη μετανάστευση. Βέβαια, οι συζητήσεις είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ελπίζω να υπάρξει κοινή θέση το στομότερο δυνατόν. Κατά την άποψή μου λοιπόν χρειαζόμαστε έναν ε, σύνολο κανόνων, ε, ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για να ξέρουμε πού πηγαίνουμε και όλα να διέπονται από τους ίδιους κανόνες. Ε, γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προγράμματα επιτόπου για τα ευρυζωνικά δίκτυα ε, από τα Ταμεία Ανάπτυξης της Υπαίθρης, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου όροι και οι δικαιώχοι, εάν θέλουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα μέσω του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής, θα πρέπει να τηρήσουν πάρα πολλούς όρους. Επομένως, πιστεύω ότι ένα σύνολο ενιών κανόνων για τα διαρθρωτικά ταμεία με ε, συγκεκριμένα κονδύλια βάσει συγκεκριμένων κανόνων θα ήταν το ιδεώδες. Ελπίζω να μπορέσουμε να είμαστε αρκετά φιλόδοξοι για το Ταμείο Οικονομικής και Δαφικής Ανάπτυξης και πιστεύω ότι αυτό θα διευκολύνει και το συντονισμό για όλες τις πηγές χρηματοδότησης. Το αυτό ισχύει και για τις διαδικασίες των ελέγχων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι προκύπτουν διάφορες ε, περιπτώσεις τις οποίες οι δικαιούχοι αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο ε, στον έλεγχο αντί της εφαρμογής. Επομένως, ε, πολύ συχνά οι διαχειριστικές αρχές και οι δικαιούχοι ε, υπόκεινται διαδοχικούς ελέγχους από διάφορες πηγές ελέγχου για την ίδια δραστηριότητα και νομίζω ότι πλέον πρέπει να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση ιδίως όταν ένας έλεγχος επιβεβαιώνει ότι όλα βαίνουν καλώς και αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Πρέπει να υπάρχει μια νέα αρχή ε, ενός ελέγχου ώστε να συντονίζονται οι διάφορες αρχές ε, στις εργασίες τους. Αυτό θα διευκολύνει και τη δουλειά όλων εκείνων που ε, εφαρμόζουν την πολιτική αυτή επιτόπου και ε, φτάνουν την Ευρώπη σε κάθε γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να σας πω ότι λυπούμε όταν βλέπω νέους ανθρώπους σε διάφορες χώρες που με λένε ότι δεν προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια γιατί οι διαδικασίες είναι μακροβόρες, ε, γραφειοκρατικές και νομίζω ότι ε, η απόδοση, η ευελιξία και η απλοποίηση θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την πολιτική συνοχή και έτσι και θα εξοπλίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και νομίζω ότι σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ΚΟΤΕΡ, με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα μπορέσουμε να δούμε πώς ε, η πολιτική συνοχή θα κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχυρότερη αλλά και πιο κοντά στις θεμελιώδεις αρχές της. Ε, ειρήνη, δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη και ευημερία για όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίτροπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτόν τον ενδιαφέροντα, για αυτήν την ενδιαφέρουσα ομιλία που νομίζω θα οδηγήσει σε πολλά σχόλια και ερωτήσεις. Όπως γνωρίζετε, έχουμε εμπειρία θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων, θα ακούσουμε τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζι, της Επιτροπής Κότερ ε, και θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Πρώτα θα δώσω όμως το λόγο στους συντονιστές ε, από την Επιτροπή Ρέτζι. Πρώτα ο κύριος Φανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να είμαστε όλοι μαζί στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Περιφερειών και Πόλεων ε, που ξεκίνησε ε, εχθές, μια συμμαχία που θέλουμε να υποστηρίξει την πολιτική, ε, την πολιτική μας. Πρέπει να υπάρξει και πολιτική πίεση. Νομίζω ότι η δική μας αίσθηση από την Επιτροπή Ρέτζη της δικής μας ομάδας είναι ότι πρέπει να δράσουμε χωρίς να περιμένουμε. Υπήρξε η έκθεση Festival, ε, η οποία ήταν πολύ συγκεκριμένη σε σχέση με αυτά που θέλουμε. Βάσει αυτή της 7ης έκθεσης για τη συνοχή γνωρίζουμε περισσότερα. Το θέμα είναι επηρεάζει άμεσα ε, τη βασική μας κατεύθυνση ε, όπως τη θέτουμε επί χάρτου για, το θέμα, ε, για τα θέματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή Ρέτζη. Η 7η Επιτροπή Συνοχής μοιάζει με την 6η και με την 5η και με όλες τις προηγούμενες γιατί ήρθε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο ήταν σαφές, ήταν γνωστό και... Ε, ε, μπορούσε κανείς να λάβει νέα μέτρα. Ε, τώρα είναι κάτι το ε, καινούριο, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι τα μέτρα και ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να κάνουμε για τη συνέχεια. Πρέπει να σκεφτούμε τους επόμενους, οκτώ τους επόμενους οκτώ μήνες. Θα περιμένουμε, θα επαναλάβουμε ξανά τα ίδια ή θα πούμε που θέλουμε να πάμε Να πούμε δηλαδή ότι το Κοινοβούλιο έχει σκοπό να, να εξετάσει όλες αυτές τις συστάσεις στη σελίδα 15, 16, 17 ε, μπορεί κανείς ε, να δει εκεί πάρα πολλές προτάσεις που προέρχονται ουσιαστικά από το έγγραφο προβληματισμού. Δεν είναι νέες ιδέες ε, σε σχέση με την συνοχή από πλευράς Κοινοβουλίου και από κοινού με την Επιτροπή Περιφερειών. Πρέπει να συμφωνήσουμε για την ταχύτητά μας, γιατί υπάρχουν ζητήματα ουσιαστικά για την πολιτική συνοχής. Ε, είμαστε αργοί σε μερικά πράγματα ε, για παράδειγμα το αποθεματικό επιδόσεων των 21 ε, δις μπορούν οι χώρες που είναι σε θέση να τα αξιοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν όπως ανέφερε και η έκθεση Φέσφαλ να περιμένουμε τι θα κάνουμε εν πάση περιπτώσει Πήγαμε προσφάτω στη Ρουμανία και είδαμε μια πολύ, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό απορρόφηση. και μπορεί να πει κανείς ότι είναι στα χέρια των κρατών μελών. Εντάξει, 400 σελίδες κανονισμοί, 200 ε, σελίδες επιπλέον για τι αποσαφηνήσει και 12.000 σελίδες για το δικαιούχο. Ε, τι κάνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που τα κάνουν όλα ένα μπάχαλο δεν θα πρέπει να επιβραβεύονται να τονίσει τρία για παράδειγμα. Τρεις, τρία χρόνια μετά από την απόφαση μπορεί να ε, υλοποιηθεί η απόφαση αυτή. Για όνομα του Θεού έχει περάσει πολύ καιρό. Έχουμε τόση εμπειρία στις πόλεις ε, για διάφορα ζητήματα ε, υπάρχει γνώση, υπάρχει ε, η συνδεσιμότητα, ε, υπάρχουν οι μεταφορές, υπάρχουν τα κοινωνικά ζητήματα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα πρέπει να φτάνουμε σε ένα σύστημα που δεν έχει αποτέλεσμα σε 7 χρόνια, αλλά θα είναι κάπως πιο ταχύ. Και συμφωνώ, περισσότερα χρήματα στο ευρωπαϊκό σκέλος, ναι, μπορούμε να δούμε η διευκόλυνση διευκόλυνση για τη ε, συνδεσιμότητα πόσο καλά λειτουργήσε. Πρέπει όμως να υπάρξει πίεση προς τα κράτη-μέλη. Αν δεν το χρησιμοποιείτε το χάσετε. Λογικό είναι αυτό. Ή απλώς δεν θα ξαναγεμίζουμε τον κορβανά. Ε, τι θα κάνουμε λοιπόν με τα χρήματα των φορολογουμένων. Το λέμε αυτό, πρέπει να το λέμε ότι δεν θα περιμένουμε, δεν θα περιμένει το Κοινοβούλιο μέχρι του χρόνου να επιληθούν κάποια από τα ζητήματα αυτά και δεν νομίζω ότι ε, υπάρχει αυτή η υποστήριξη. Το Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει δράση. Και κάτι ακόμη, μία πρώτη παρατήρηση από πλευρά μου. Χθε, ε, στη συνεδρίαση των συντονιστών, συζητήσαμε για την ταχύτητα που θα θέλαμε να έχουμε. Ο συνάδελφο εδώ που κάθεται δίπλα μου θα δουλέψει μαζί μου για αυτή την έκθεση, για αυτή την 7η έκθεση συνοχή από πλευρά Επιτροπή ε, Περιφερειών. Μία παρατήρηση θα ήθελα να κάνω, γιατί προσπαθώ να είμαι σύντομος. Ε, δύο εκθέσεις μας ε, της ΚΟΤΕΡ που αφορά το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής μετά από το 2020 και αφορά την απλοποίηση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Σας το λέω, μπορείτε να τη βρείτε στο βάθος της αίθουσας. Συντονιστής του ΕΛΚ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, από την 7η έκθεση για τη συνοχή Διαφαίνεται ότι υπάρχει οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη, αυξάνεται το ΑΕΠ, αυξάνεται και η απασχόληση. οι περιφερειακές ε, διαφορές μειώνονται, όχι όμως παντού. Και το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο αυτό είναι παρκές. Εγώ προέρχομαι από τη Σλοβενία. Πρέπει να πω ότι οι πολίτες μας δεν ε, έχουν τη βεβαιότητα, δεν έχουν βεβαιότητα για το μέλλον τους, έχουν πολλές ανησυχίες και πολλές ανασφάλειες και στις περιφέρειες ε, τις πιο μακρινές αυτό είναι ακόμη εντονότερο. Πρέπει αυτή τη στιγμή και επί τη βάση αυτής της έκθεσης να μιλήσουμε για την πολιτική συνοχή του μέλλοντος μετά το 2020. Κατά τη γνώμη μου χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη πολιτική συνοχή, ε, μεγαλύτερη επικουρικότητα, απλούστευση, ε, ευελιξία και αλληλεγγύη. Το πολιτικό όραμα της ε, Επιτροπής Περιφερειών αναφέρθηκε στη γνωμοδότηση τους, ε, του Μίχαηλ Σνάιντερ, μια γνωμοδότηση αυτής της χρονιάς ανεξαρτήτως ε, των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να συζητηθεί το οικονομικό πλαίσιο που θα υποστηρίξει την πολιτική συνοχής στον ίδιο βαθμό όπως και τώρα. Πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι ανάγκες των πολιτών μας ε, και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να καταλάβουν, να νιώσουν τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ ε, με τη συμμαχία, τον συντονισμό για την ε, συνοχή. Είμαι υπέρ ε, του να είναι η πολιτική συνοχή σε μία από τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς όσους έχουν ε, επεξεργαστεί την πολιτική αυτή και έχουν δουλέψει για αυτήν, προς την κυρία ε, Κρέντου το λέω αυτό, προς τον Επίτροπο Έτιγκερ. Ευχαριστώ και όλους τους ευρωβουλευτές. Επιτρέψτε μου να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω ε, τη Βουλγαρική Προεδρία για την εκδήλωση που θα γίνει το 2018 στη Σόφια πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για την αποτελεσματικότητα της εδαφικής συνοχής ε, στο μέλλον. Ε, Κάποιες πρώτες σκέψεις. Η έκθεση μόλις εχθές παρουσιάστηκε και σήμερα γίνεται μια πρώτη συζήτηση άλλωστε. ένα γενικό όρο με τον οποίο συμφωνώ. Αυτή τη στιγμή βγαίνουμε από μία από τις πιο οξύες και φρικτές οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις που βίωσε η Ευρώπη στο πρόσφατο παρελθόν. Και επομένως καλό είναι να δούμε πώς ε, η πολιτική συνοχής ε, λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια. Τι ε, αντίκτυπο είχε, κυρίως για να αποφύγουμε να αμβληθούν οι αποστάσεις μεταξύ των περιφερειακών συστημάτων. Και αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται διότι στην ολοκλήρωση αυτού του κύκλου βλέπουμε ότι οι συνέπειες της κρίσης ε, και η έξοδος από την κρίση ε, είναι τελείως διαφορετικά. Αλλιώς ε, τα βιώνουμε στη Βόρεια Ευρώπη, αλλιώς στη Νότια, αλλιώς στην Ανατολή, αλλιώς στη Δύση. Και εδώ υπάρχει ένας πολύ ουσιαστικός λόγος να ενισχύσουμε την πολιτική συνοχής. Να υπάρχει μια διάσταση η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των ευρωπαϊκών περιφερειών, αλλά να υπάρχει και μια πολιτική συνοχής η οποία ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει και το λόγο ύπαρξή τη, να μειώσει τις αποστάσεις μεταξύ των περιφερειών και να συνοδέψει τις διάφορες διαδικασίες σύγκληση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πρώτο σημείο στο οποίο θα πρέπει να επιμείνουμε, προκειμένου να βρούμε και τους λόγους ε, για τους οποίους θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα ε, για την πολιτική συνοχή και να συνοδεύσουμε τα επόμενα χρόνια και με χρηματοδότηση αλλά και με πολιτικές αυτή την πολύ ε, ουσιώδη πολιτική που χαρακτήρισε την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο ζήτημα, και εδώ συμφωνώ και με την παρατήρηση του συναδέλφου Φανίστερ Λόι, αυτή τη στιγμή μας απομένουν 8 μήνες μέχρι να υποβληθεί και το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της πολιτικής συνοχής αλλά και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, τι θα κάνουμε σε αυτό το οκτάμινο. Τι εργασίες θα πρέπει να κάνει κυρίως η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σε στενή σχέση με τους συναδέλφους και φίλους από τα άλλα ε, θεσμικά όργανα, κυρίως την Επιτροπή των Περιφερειών, ώστε να συνοδέψουμε τις αποφάσεις οι οποίες από εκεί και πέρα ε, θα οριστικοποιηθούν ε, μέσω της παρουσίασης της έκθεσης. Το θέμα της απορρόφησης, για παράδειγμα, θα μας απασχολήσει. και θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας και να προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μαζί, κυρίως με τους αδέλφους της Επιτροπής Κοτέρ, να δούμε ε, ποια ε, ήταν τα αίτια των αποστάσεων. Η ευρωπαϊκές ε, προκλήσεις ήταν αυτές οι οποίες ε, δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα και είναι τελείως διαφορετική η εφαρμογή. Πολύ συχνά οι διάφορες περιφέρειες ε, αντιμετωπίζουν πρόβλημα να τηρήσουν το σύμφωνο σταθερότητας της δημόσιας επενδύσεις. Υπάρχει πρόβλημα με το διοικητικό μηχανισμό, πώς θα μεταρρυθμεί στη ο διοικητικός μηχανισμός. Εγώ πιστεύω ότι στο θέμα της απορρόφησης δεν θα πρέπει να είναι ουσιαστικά η ασπίδα βάσει της οποίας θα πούμε ναι ή όχι στην πολιτική συνοχή. οσο η Επιτροπή ρετζη και Κοτέρ θα πρέπει να συνεργαστούμε το επόμενο οκτάμινο για να βρούμε και να διευκρινίσουμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έκαναν πιο περίπλοκη την αυπορόφηση σε αυτό το στάδιο και γιατί προέκυψε αυτό το πρόβλημα σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες περιφέρειες και γιατί σε κάποιες άλλες ήταν πολύ πιο εύκολη διαδικασία. Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία τα οποία επέτρεψαν ε, ε την επιτυχία της πολιτικής συνοχής. Ε, νομίζω ότι εδώ θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το θέμα λίγο περαιτέρω. Και δύο τελευταίες παρατηρήσεις και με αυτές ολοκλήρωσα γιατί αλλιώς θα χάσουμε πολύ χρόνο. Το ένα αφορά τη σχέση ε, με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είναι απόλυτα προφανές ότι μια πολιτική με 7 χρόνια προγραμματισμού και εξέλιξης δεν μπορεί να δοκιμάζεται κάθε φορά στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Επομένως, πρέπει να αποφασίσουμε τι σχέση πρέπει να υπάρχει μεταξύ πολιτικής συνοχής και της οικονομικής διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Και κατά με εδώ υπάρχει κάτι το οποίο αφορά κυρίως ε, την ε, ε, ανάκαμψη των δημοσίων επενδύσεων και τη μεταρρύθμιση του διοικητικού μηχανισμού. Νομίζω ότι στα δύο αυτά σημεία θα μπορούσαμε να ζητήσουμε βοήθεια ε, από καιρού καιρών ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να δημιουργήσουμε μια κάποια σχέση. Βλέπω ότι δεν τίθεται εκ νέου το θέμα τη μακροαιρεσιμότητα, διότι διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν ανεφάρμοστα. Ελπίζω να το έχουμε αφήσει πίσω μα αυτό το θέμα και να μην ξαναεμφανιστεί στου νέου κανονισμού. Όπω και να έχει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό ήταν ένα θέμα και από θεωρητική σκοπιά κατά την άποψή μου λανθασμένο. Λανθασμένα αντιμετωπίστηκε και εφαρμόστηκε και αποδείχθηκε αυτό και με τα όλα θέματα που αφορούσαν την Ισπανία και την Πορτογαλία πόσο δύσκολο ήταν να εφαρμοστεί. Τέλος, συμφωνώ για το ενίο ταμείο. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο μεταρρύθμισης και απλοποίησης και θα ήθελα να επιμείνω πάρα πολύ σε αυτή την πτυχή διότι ε, αυτό ε, θα έδινε και τη δυνατότητα από τη μία προγραμματική περίοδο στην άλλη να γίνει μια μετάβαση πολύ πιο γρήγορη. Αυτό που χρειαζόμαστε δηλαδή. Ε, έχουμε 8 μήνες εντατικών εργασιών, συνεργασιών, αντιπαράθεσης για να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική συνοχή στα επόμενα χρόνια. ευχαριστώ. Τώρα, να ακούσουμε από την πλευρά της Κοτέρα τον συνάδελφο. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι και σύντομος. Αυτή η έκθεση, η έκθεση για τη συνοχή, προβλέπει το τι θέλει να κάνει και προτίθεται να διακηρύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς επίσης ότι η πολιτική συνοχή λειτουργεί βασικά αν ε, προσμετρηθούν δείκτες ε, για την ε, απασχόληση, για το ΑΕΠ κατά κεφαλή, η πολιτική συνοχή λειτουργεί ως μέτρο. Ένα ενδιαφέρον θέμα για μένα είναι πώς θα αισθανόσασταν αν δεν είχε υπάρξει η πρώτη, δεύτερη έως και έβδομη έκθεση συνοχής προηγουμένως. Νομίζω ότι το αίσθημα που επικρατεί είναι ότι τα πράγματα αυτά είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ισχύουν τώρα το 2017. Και αυτό πάλι αποτυπώνει ότι λειτουργεί η πολιτική συνοχή. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε ενδεχομένω στο σημείο αυτό είναι ότι οι περιφερειακές, ή μάλλον εδαφικές προοπτικές ε, και πτυχές της πολιτικής συνοχής δεν είναι καλά προσαρμοσμένες. Στο κεφάλαιο για την ε, εδαφική συνοχή δεν υπάρχει λεπτομερής ανάλυση των ε, εδαφικών προκλήσεων και αυτό είναι ατυχές πιστεύω. Η πολιτική συνοχή αποτελεί απλώς μία πολιτική αυτό που είναι σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το τι κρύβεται πίσω από την πολιτική αυτή. Τα εργαλεία, τα μέσα που μας επιτρέπουν την υλοποίηση της πολιτικής. Και δεν εννοώ α, με τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και να κοιτάξουμε την εδαφική πτυχή της συνοχής, θα πρέπει να το κάνουμε αυτό και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό, το τομεακό, δημόσιο και τοπικό επίπεδο. Η ενοποιημένη λοιπόν εδαφική πτυχή της πολιτικής συνοχής είναι κάτι το οποίο, στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε πιο πολύ προσοχή από ότι έως τώρα η πολιτική συνοχή λειτουργεί, αλλά θα πρέπει να της δώσουμε και την εδαφική και την ενοποιημένη διάσταση την οποία δεν έχει στην παρούσα φάση. Σα ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητή από την ε, Ρέτζη, η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επιτροπέ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την ομιλία σας και υποστηρίζω την έκθεσή σας και όλους διτέρου του Πετροπυλώνα. Πιστεύω ότι θα συνεπάγεται αυτό μεγαλύτερη δαπάνη ε, εξόδων. Επίση, πιστεύω ότι οι μελλοντικέ δομέ θα είναι καθοριστική σημασία. Είπατε ότι αυτό βρίσκεται προ συζήτηση στην παρούσα φάση και αυτό αναπτύσσεται. Μπορούμε να συζητήσουμε με λεπτομέρεια τις ε, διαρθρωτικές αυτές μεταρρυθμίσεις, αλλά όποτε συζητάμε τέτοια ζητήματα, εγώ πάντα ζητώ λεπτομέρειες. Θα μπορούσατε να μας δώσετε πιο πολλές λεπτομέρειες. Ευχαριστώ από την Κοτέ, κύριε Φανερμαϊρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση για την πολιτική συνοχή έρχεται σε ένα πάρα πολύ κέριο χρονικό σημείο, γιατί μπορεί να αποτελέσει, αν θέλετε, τη βάση για τη μελλοντική πολιτική συνοχή. Σύμφωνο με το σημείο που έθιξε ο κ. Φανίστελ Ρόι, τόνισε ότι θα πρέπει τώρα να δράσουμε, να διατηρήσουμε αυτή την ορμή που έχει δημιουργηθεί και νομίζω ότι πολλές έρευνες και μελετές καταδεικνύουν ότι υπάρχουν ουσιαστικά αποτελέσματα στην ε, πολιτική συνοχή. Ωστόσο, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πιο πολλά. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι μόνο, όχι μόνο η εδαφική συνοχή, <coughs> αλλά προστιθέμενη αξία για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, εθίχθη ένα θέμα το οποίο έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Πώς θα περιγράψουμε τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Έχουμε μεγάλα διαφορές. στη Σουηδία, για παράδειγμα. Έχουμε 40 διαφορετικούς ορισμούς σε ό,τι αφορά τις περιοχές, τις περιφέρειες. Έχουμε περιοχές όπου είναι υψηλή η ενέργεια, το προσδόκιμο είναι χαμηλότερο ή υψηλότερο. Υπάρχουν πολλές λοιπόν τέτοιες διαφορές και δεν βλέπουμε τέτοια στατιστικά στοιχεία. Υπάρχουν ε, περιοχές ε, στην Ήπεθρο όπου είναι ανησυχητική η γύρανση του πληθυσμού. Χρειαζόμαστε λοιπόν τέτοια στοιχεία και τέτοια δεδομένα για να γίνει σωστή ανάλυση των προκλήσεων με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πιο εξειδικευμένες πληροφορίες. από το εθνικό επίπεδο, αν θέλετε, από τα μέσα προς τα έξω, τα πράγματα φαίνεται πηγαίνουν καλά, αλλά χρειαζόμαστε μια συνολική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά και την βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε απέναντί μας. ένα στοιχείο λοιπόν είναι σαφέ στην έκθεση αυτή. Για πρώτη φορά στην Ευρώπη έχουμε όχι πολλά άτομα που πεθαίνουν από τη καινούργια άτομα που γεννιούνται. Αν θέλουμε λοιπόν ένα σύστημα πρόνοια στην ε, κοινωνία μας, χρειαζόμαστε ανανέωση του πληθυσμού, χρειαζόμαστε πιο πολλά άτομα να εργάζονται για να χρηματοδοτούν το πρόγραμμα αυτό. Έχουμε συζητήσει και το θέμα των γυναικών και την απασχόληση των γυναικών και την απασχόληση των πρεσβυτέρων. Έχουμε και το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο επίσης ε, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ε, ενσωμάτωσης των ασύλων άσυλο και το πώς θα συνεισφέρουν στα συστήματα πρόνοιας. Οι εκθέσεις λοιπόν αυτές ε, καταδεικνύουν ότι όταν συνδέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και εξετάσουμε το πώς μπορούμε να δώσουμε πρόσβαση στην παλαιότερη γενιά σε αυριζονικότητα και το καθεξής. Αυτό είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει στην Σουηδία. Έχουμε εργαστεί πολύ για θέματα προσβασιμότητας σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα μέσα συγκοινωνίας για τις ε, πρεσβύτερες γενιές. Ακόμα και αν αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας, θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα νέα ζητήματα να αντιμετωπιστούν στην πολιτική συνοχή. Και με τον τρόπο λοιπόν αυτό πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κ. Φαμίλτον Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Επιτροπή, πάντα με χαρά σα υποδεχόμαστε εδώ στην Επιτροπή μα. Και ακόμα μεγαλύτερη χαρά που έχουμε εκπροσώπου τη επιτροπή των Περιφερειών εδώ στην αίθουσα. Από όλη την Ευρώπη. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη που καθυστέρησα στην αφήξή μου και δεν άκουσα το πρώτο κομμάτι της εισαγωγής σας. Με ε, ενημέρωσαν ως μέλος ε, από την Ολλανδία για το νέο συνασπισμό, κυβερνητικό συνασπισμό που σχηματίστηκε στην Ολλανδία. Χαίρομαι μεν, από την άλλη στενοχωριέμαι και λίγο, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ Βέλγων και Ολλανδών. Δεν σπάσαμε το παγκόσμιο ρεκόρ για τη δημιουργία λοιπόν ε, κυβέρνηση, του σχηματισμού κυβέρνηση. Να δούμε, λοιπόν. Mm-hmm. Αλλά -hmm. Αλλά σοβαρευτούμε. Έβδομη έκθεση για τη συνοχή. Χαίρομαι που σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση εστιάσατε πιο πολύ στο θέμα της υπέρβαση των εμποδίων σε όλα στις ευρωπαϊκές χώρες, πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα δηλαδή. Και εγώ και η ομάδα μου είμαστε υπέρ του ίντερ και για το μέλλον. Αυτό επιτρέπει πιο πολλές επενδύσεις στις μεταφορές, στις υποδομές, σε απόμακρες περιοχές, επενδύσεις σε κοινά κέντρα ερευνών σε όλη την Ευρώπη. Συμπεριλεχθεί και αυτό και στην έκθεση ΒΕΣΠΑ και επίσης ε, έτσι δίνονται ευκαιρίες και σε χρηματοδότηση και επενδύσεων. ο διάδοχο αν θέλετε του Interreg Europe πρόγραμμα. Έρευνα, καινοτομία, ανάπτυξη, οι περιβαλλοντικέ προκλήσει, όλα αυτά δεν γνωρίζουν ευρωπαϊκά σύνορα. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε από κοινού σε όλη την Ευρώπη. Επίση, αυτό αφορά και τι επενδύσει στον κόσμο, γιατί θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία του Interreg στην διασυνοριακή συνεργασία και σε ό,τι αφορά τη βελτίωση τη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού πέρα από τα κρατικά σύνορα. Χαίρομαι λοιπόν που εστιάζεται στο θέμα αυτό. Δεύτερο ζήτημα, οι αστικές πολιτικές συνοχής. Έχουμε το καινοτομικό αυτό πρόγραμμα το οποίο και επεκτάθηκε και χαίρομαι για να συμπεριλάβει και χρηματοδότηση και προγραμμάτων ε, καινοτόμων σε όλες τις πόλεις, γιατί οι πόλεις είναι κινητήριε δυνάμεις, αν θέλετε, της Ευρώπης ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συνέχεια και μετά το 2020. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει mainstreaming. Θα πρέπει να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των πόλεων σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση μπορεί να είναι οικονομικά μέσα αλλά και κλασικές επιδοτήσεις. Επίσης να δούμε τι θα έχει ως αποτέλεσμα το, το σύμφωνο του Άμστερνταμ με τις θεματικές ενότητες του για να πραγματικά να υποφεληθούμε από αυτή την ορμή που έχει δημιουργηθεί στην πολιτική συνοχή. θα σα ακουστεί υπερβολικό αυτό, αλλά νομίζω ότι για τι πόλει τη Ευρώπη και για την Ευρώπη ε, διακυβεύονται πολλά. Τρίτο σημείο, θα υπάρξουν νέε δημοφιλικέ προτάσει, θα υπάρξει ένα νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και χαίρομαι με την ομάδα μου που δεν υπάρχει επανάσταση, αλλά εξέλιξη, αν θέλετε, μεταξέλιξη της πολιτικής συνοχής. Πολιτική συνοχή 2.0. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ε, βελτιώσεις, παρά το γεγονός ότι πολλοί από εμά θα θεωρήσουν ότι μετά το 2020 θα έχουμε πιο πολλά χρήματα για να εκπληρώσουμε πιο πολλούς στόχους. Αυτό όμως είναι ε, η πραγματικότητα. Άρα θα πρέπει να κάνουμε πιο πολλά σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά μας μέσα, τα τα μέσα ανα, ανακύκλωσης, revolving funds. Θα πρέπει να δούμε και ποιος είναι, ποια είναι η σύνδεση μεταξύ των συστάσεων αναχώρα, τα ευρωπαϊκά εξάμεινα και την πολιτική επενδύσεων. Και θα πρέπει να επικεντρωθούμε πιο πολύ σε μικρομεσαίες επιχειρήσει στην καινοτομία, αλλά και στο να καταστεί η ευρωπαϊκή πολιτική πιο ανθεκτική σε ό,τι αφορά και την αλλαγή του κλίματο μεταξύ άλλων. Αν ενισχύσουμε την πολιτική συνοχή με τον τρόπο αυτό, νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα προσπιστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κριτική του κόσμου που πάντα α, βάλει κατά της πολιτικής ε, συνοχής. Εμείς ε, από την άλλη και νομίζω ότι μιλώ και εξ ονόματος της Πρόεδρου με αυτόν τον τρόπο εργαζόμαστε και θα σας χορηγήσουμε ένα έγγραφο τοποθετήσεις με την ε, άποψη και τοποθετήση των φιλελευθέρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας για να πετύχουμε ένα και μόνο πράγμα να υπάρξει αυτή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία την οποία όλοι επιδιώκουμε. Ευχαριστώ. Από την Κοτέρ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Ρέτζη. Χαίρομαι ιδιαίτερος που είμαι εδώ πάλι. Νομίζω πολλοί από τους προλαλήσεις είπε, είπαν ότι πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα, όπως για παράδειγμα το κεφάλαιο 6 που είναι μια ιστορία επιτυχίας αποκρισταλώνει τη δουλειά που έχει γίνει. Αν το προσθέσουμε αυτό στο highlights document ε, και έπρεπε να διαλέξουμε τι, αν θα κρατήσουμε την πολιτική συνοχή ή όχι, νομίζω ότι το κεφάλαιο 6, το έγγραφο highlights και γενικώ ολόκληρο το έγγραφο ε, είναι πάρα πολύ ισχυρό πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ Κότερ και Ρέτζι και εγώ θα ήθελα να υπάρξει μία συνεργασία όσον αφορά ε, τις ε, βασικές, ε, τα βασικά βήματα που θα ακολουθήσουμε. Ε, πρέπει να δημοσιεύσουμε πολύ περισσότερο τις επιτυχημένες ιστορίες της πολιτικής συνοχής και όταν βλέπω συνεχώς τη λέξη κρίση στο έγγραφο, εντάξει υπάρχουν πολλές προκλήσεις αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που ως μέλος της Επιτροπής Κότερ πηγαίνω σε διάφορες πόλεις κάθε εβδομάδα και με ρωτούν Λοιπόν όλοι αν είμαστε, προς, ε, αν είμαστε στο σωστό δρόμο. Πραγματικά θεωρώ ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και τα πράγματα πηγαίνουν καλά και συμφωνώ με τη λέξη εξέλιξη ε, που χρησιμοποίησε ο κύριος Φαν ε, νομίζω ότι είναι ε, εξέλιξη και όχι επανάσταση. Πρέπει να υπάρχει λίγο περισσότερη επικοινωνία, πρέπει ε, λίγο περισσότερο να έχουν την ευκαιρία οι επόμενες γενναίες να δουν τις περιφέρειές τους, να γίνουν οι φάροι της εξέλιξης και της πρόοδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε τη σημασία σημασία της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειαζόμαστε μια καλύτερη και δυνατότερη σχέση εργασίας. Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει επαρκής αναφορά στην Επιτροπή ε, Περιφερειών ε, στην 7η έκθεση της πολιτικής συνοχής, γιατί Κάθε περιφέρεια έχει δώσει πληροφορίες ε, στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής. Έχουν υπάρξει τόσες πολλές γνωμοδοτήσεις από πλευράς μας ε, όσον αφορά τη βελτιωμένη, τους βελτιωμένους δείκτες ε, για την εδαφική συνοχή και δεν θεωρώ ότι έχει επαρκώς αντικατοπτριστεί στην έκθεση. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εντύπωση. Πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο. Ε, θα μ' άρεσε πάρα πολύ λοιπόν να γίνει μια παρουσίαση για αυτά τα building blocks, να δούμε ε, τι μπορούμε να κάνουμε, να μην χάνουμε το χρόνο μας, να ε, συναντιόμαστε δύο φορές το χρόνο κατά αυτόν τον τρόπο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την πολιτική συνοχή. ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση και συμφωνώ με τον κύριο Φανίστελρο ότι πρέπει να δράσουμε τώρα και να μην περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ η κυρία ε, Μισελς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε πρόεδρε ίσως, ως πρώην μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών και ενεργό μέλος εδώ της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαίρομαι που υποδεχόμαστε εδώ τους συναδέλφου τους οποίους ε, γνωρίζω και δεν γνωρίζω, τον κύριο Μπορ, τον οποίο γνωρίζω από παλιά, για παράδειγμα, χαίρομαι που η συνεργασία μας έχει προωθηθεί σε ό,τι αφορά την εξέλιξη ή την επανάσταση. Evolution ή revolution. Δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά να πω το εξή ε, προς ε, την Άλτε, ότι το σημαντικό είναι να μην μείνουν τα πράγματα εκεί που βρίσκονται σήμερα. Τώρα, αν θέλετε να το πείτε evolution, revolution, ό,τι θέλετε πείτε το. Εξέλιξη ή επανάσταση. Η έβδομη έκθεση για τη συνοχή λοιπόν μου προκάλεσε εν μέρη θετικές εκπλήξεις. Η σαφήνεια της διαπίστωσης, για παράδειγμα, ότι το χάσμα μεταξύ των φτωχών και πλούσιων περιφερειών έχει οξυνθεί. Μου προκαλεί έκπληξη. Αλλά αυτό που μου προκαλεί θετική έκπληξη είναι ότι υπάρχουν σαφείς προσανατολισμοί σε ό,τι αφορά το πόσο απαραίτητη είναι η πολιτική συνοχής. όλοι όσοι συμμετείχαν στις συζητήσεις τις τελευταίες μήνες ξέρουν ότι αυτό δεν είναι δεδομένο να μπει αυτό ως δήλωση δηλαδή. Ευχαριστούμε λοιπόν την κυρία Κρέτσου για τα ξεκάθαρα αυτά λόγια. Στατικό επίσης είναι ότι υπάρχει σαφής ε, αναφορά στις μεταβατικές περιφέρειες. Να δούμε λοιπόν και στην πολιτική συνοχή κατά πόσον χρειάζεται. Αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά αποτελούν σωστές προσεγγίσεις. Και πιστεύω ότι η κυρία Κρέτσου, η κυρία Επίτροπος προηγουμένως ε, ανέφερε τα βασικά, τα σωστά βασικά ζητήματα. Τώρα βέβαια να περάσω και στο αλλά. αλλά. Αυτά που είπε ο κύριος Φανίστεροι. Θα τον εκπλήξω ενδεχομένω. Πιστεύω ότι η έκθεση παρόλα αυτά δεν έχει επαρκείς συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είμαστε στο πρώτο έτος ε, της συζήτησης για το πώς θα αναπτυχθεί περαιτέρω η πολιτική συνοχή. Η Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αμφότερα τα όργανα, έχουν υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις. Θα ήθελα λοιπόν στην 7η έκθεση για τη συνοχή κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που ανέφερε και ο Άλμπερτ Μπόρ για τις εδαφικές προκλήσεις για παράδειγμα, την εδαφική πτυχή για το πώς ε, και ποια συγκεκριμένα μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ποια μοντέλα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Εδώ θα ήθελα λίγο παραπάνω τόλμη, λίγο παραπάνω θάρρο στη συζήτηση για να μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά υποστηρίζουμε και προσπιζόμαστε την πολιτική συνοχή και εκ παραλλήλου μία μεταρρύθμιση στο πλαίσιο των τρέχουσων μεταρρυθμίσεων δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποφύγουμε. Άρα, αφενός έχω να πω ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία, από την άλλη όμως ε, θα πρέπει σίγουρα τους επόμενους οκτώ μήνες να κάνουμε μια πιο συγκεκριμένη προτάση. Ιδάλλως θεωρώ ότι θα έχουν δίκιο να συνεχίσουν την κριτική όσοι μας επικρίνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και Πρόεδρος. Uh, Καλημέρα, κυρία Μιχαήλοβα, κυρία Κρέτσου, κύριε Όσφαλτ, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα επικεντρωθώ σε μία πτυχή στην οποία επικεντρώνομαι πάντα, η διασυνοριακή συνεργασία. Και θα ήθελα να συμπληρώσω αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο που επετεύχθη. Στην έκθεση, έκθεση υπήρχαν δύο ε, παράγραφοι που λένε ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία. Τώρα υπάρχει μια πιο εις βάθος ανάλυση και νομίζω ότι το όλο θέμα της αναθεώρησης των διασυνοριακών θεμάτων είναι επιτυχία. Ήταν, ε, υπήρξε μια επιστημονική συστηματική προσέγγιση για την ανάλυση ε, των συνοριακών φραγμών που εξακολουθούν να υπάρχουν. Και το αποτέλεσμα είναι ότι επιτέλους έχουμε ένα αριθμητικό στοιχείο. Ένα αριθμητικό στοιχείο που συνδέει τις επενδύσεις ε, με την ε, ανάπτυξη του ΑΕΠ όταν ε, ξεπερνιούνται τα εμπόδια αυτά. Και Εάν άρουμε τα εμπόδια που υπάρχουν ακόμα στα σύνορα, μπορούμε να έχουμε και 2% αύξηση. Ε, και ως οικονομολόγος να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό το στοιχείο, πολύ μεγάλος αριθμός, δεν είναι μηδαμινό και ε, πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις για να άρουμε τα ε, εμπόδια στα σύνορα και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε επενδύσεις. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η διασυνοριακή συνεργασία υπερβαίνει την οικονομική ανάπτυξη. Εγώ ζω σε ένα μικρό χωριό και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ε, πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να υπάρξει στην ποιότητα ζωής όταν έχεις ένα καλό γείτονα ή ένα δύσκολο γείτονα. Ε, και εμείς αναφερόμαστε πάντα στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Αν επενδύσουμε λοιπόν πέραν στην οικονομική ανάπτυξη, στις ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των συνόρων, ε, προγράμματα μεταξύ ε, ατόμων μπορεί να βελτιώσει τη συνοριακή ζωή τα άτομα που ζουν στις μεθοριακές περιοχές. Αυτά λοιπόν, ε, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Βάνα. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επίτροπο ήρθε και πάλι στην Επιτροπή μας για να συζητήσουμε, γιατί η πολιτική συνοχή, η 7 πολιτική, έκθεση για την πολιτική συνοχή ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε με μεγάλη ανυπομονησία. Θα ήθελα λοιπόν να κοιτάξω από πλευρά των πρασίνων ποια ζητήματα μας απασχολούν ιδιαίτερω για την επόμενη περίοδο. Καταρχάς, θα συμφωνήσω με την προλαλή σα, με τη συνάδελφα από την ΚΟΕ. Θα ήθελα καταρχάς να βάλω μια θετική χρειά για πολλές αλλαγές που έγιναν από την ε, έκτη έκθεση. Πολλά ζητήματα τα οποία είναι ένα απόσπαστο σύστημα, στοιχείο της ε, πολιτικής για τη συνοχή σε ό,τι αφορά και τις δημόσιες επενδύσεις. Σε κάποιες περιοχές και περιφέρειες ε, τα μία ταμεία είναι οι μοναδικές δημόσιες επενδύσεις και πιστεύω λοιπόν ότι και το οικονομικό σκέλος αλλά και οι κοινωνικές επιπτώσεις της πολιτικής συνοχής είναι τεράστιες και δεδομένου και των όσων είπατε, θα συμφωνήσω ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις στοχευμένες, στοχευμένες στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν και τη βάση για τη χρήση των τριφωτικών ταμείων. Αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τους στόχους του 2020. Μία πρώτη ερώτηση λοιπόν κυρία Επιτροπέ, το δείξατε και ως μία βασική πρόκληση και η έκθεση για τη συνοχή είναι σαφέσταστη. Τα μέτρα για την προστασία του κλίματος εδώ είναι δεδομένο ότι μένουμε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με το στόχο που είχαμε θέσει. Το αποφάνθηκε σχετικά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το 20% ως δαπάνες για μέτρα προστασία ε, του κλίματος ε, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επιτευχθεί ο στόχος. Και παρά το γεγονός ότι γίνονται πάρα πολλές ε, καλές προσπάθειες και υπάρχει καλή θέληση αυτό που το αμφιλεγούμε, και εγώ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαπιστώνουμε ότι λείπουν βασικές υποδομές, ε, post-tracking και μια διαδικασία υποπτίας. Ρωτώ λοιπόν, σε ό,τι αφορά το στόχο της προστασίας του κλίματος. Εδώ χρειαζόμαστε σαφείς ε, πρόοδους για να πετύχουμε τους στόχους μας. Πώς λοιπόν θέλετε να πετύχετε το 20% των δαπανών για μέτρα προστασίας του κλίματος και την τρέχουσα περίοδο αλλά και την επόμενη περίοδο και σε ό,τι αφορά τους στόχους του ΣΚΟΠ 21 να καταστούν πιο φιλόδοξοι γιατί νομίζω ότι ε, δεδομένης και της αποχώρησης των ΗΠΑ εμείς θα πρέπει ακόμα πιο εντατικά να ακολουθήσουμε τους στόχους μας. Μια δεύτερη ερώτηση. Ανάπτυξη νέων δίκτων. Νέοι δίκτες. Ένα θέμα το οποίο θίγω σε κάθε περίοδο. Στην έκτη έκθεση είχατε ανακοινώσει ότι θα αναπτυχθούν και άλλοι δείκτες για τις επενδύσεις πέρα από το ΑΕΠ. Ότι πρόκειται λοιπόν να αναπτυχθούν νέοι δείκτες. Δεν βλέπω όμως την 7η έκθεση να υπάρχει κάτι τέτοιο. Λείπει αυτό. Απουσιάζει. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει και άλλους δείκτες, για παράδειγμα περιβαλλοντικούς δείκτες, δείκτες αναδιατομής και άλλους δείκτες που έχουν καταρτήσει οι εμπειρογνώμονες και που θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ χρήσιμοι στην περιφερειακή πολιτική. Τελευταία ερώτηση. Δείξατε ένα από τους πιο βασικούς στόχους, στην καταπολέμηση της ανεργίας και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ερωτώ. Το ESF Share δηλαδή το μερίδιο του κοινωνικού ταμείου στα κράτη-μέλη. Μήπως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση για την ανεργία. Μήπως θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό 13% για παράδειγμα και να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής του κοινωνικού ταμείου σε ό,τι αφορά τις περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερως από ανεργία για να αντιμετωπιστούν οι αδικίες και οι ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών. Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κοτέρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι σίγουρος ότι με τον νέο πρόεδρο της Επιτροπής Κότερ η δουλειά μας θα πάει ακόμη καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Τα πορίσματα της 7ης έκθεσης για την πολιτική συνοχή ε, είναι κατά τη γνώμη μου ότι η πολιτική συνοχής ε, λειτουργεί και διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη ε, και τις επενδύσεις. Αν δει ε, το γράφημα της σελίδας 185, οι συνέπειες ε, της πολιτικής συνοχής στο ενωσιακό ΑΕΠ είναι πάρα πολύ καλές και υπάρχει και ένα αριθμητικό στοιχείο στη σελίδα 22. Υπάρχουν λοιπόν αριθμητικά στοιχεία που μας, που μας δείχνουν εμ ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες ε, η πολιτική συνοχής ε, εκπροσωπεί ε, άνω του 80% των επενδύσεων. Παρά το γεγονός λοιπόν της σημασίας της κοινή μας συνεργασίας υπάρχει περίεργο κλίμα και μια επικίνδυνη κατάσταση. Οπότε θα ήθελα να σας κάνω μια βασική ερώτηση, βασική κατά την άποψή μου. Ε, οι περιφερειακές αρχές και η πολιτική συνοχή υφίστανται επίθεση ή όχι. Ποια είναι η δική σας άποψη, γιατί εμένα μου φαίνεται ότι η συνοχή αυτή τη στιγμή υφίσταται επίθεση και θα ήθελα να είμαι σαφέστερος ε, κάνοντας τρεις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση διατηρούμε για το μέλλον το ίδιο επίπεδο πόρων ε, και χρηματοδότησης ε, στην ε, προγραμματική περίοδο μετά το 2020 σε σχέση με το παρελθόν ή όχι. Γιατί, κοιτάξτε, η πολιτική συνοχή χωρίς καθόλου χρηματοδότηση δεν, δεν, δεν, αποτε, δεν, δεν, δεν είναι τίποτα. Επίσης, αυτό που αναφέρεται σελίδα 179 της έκθεσης, Υπάρχει μια θετική αξιολόγηση σε σχέση με τις εκ των προτέρων ερεσιμότητες ε, στο κεφάλαιο που μιλά για τις προτάσεις βελτίωσης ε, ε, της πολιτικής συνοχής. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε, θα μπορούσαν αυτές οι αιρεσιμότητες να εισαγάγουν το κίνδυνο ε, κάποιο χρηματοδότησης ε, που δεν θα είναι διαθέσιμη για όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό η πολιτική συνοχή να είναι ένα εργαλείο για όλες τις περιφέρειες και όχι για κάποιες. Εγώ προτιμώ την άλλη πρόταση να, ε, στο, να είμαστε περισσότερο επικεντρωμένοι στα αποτελέσματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα υπάρχει περίπτωση να εισαγάγει αυτό το κίνδυνο μιας προτιμησιακής μεταχείρισης για να το πω έτσι. Σελίδα 168 της ε, έκθεσης ε, αναφέρεται ότι το επίπεδο των δημοσίων επενδύσεων μειώνεται και είναι πολύ πιο ε, κεντρικό από το παρελθόν σε σχέση με την αποκέντρωση των δημοσίων επενδύσεων, η οποία μειώνεται συνεχώς. Για μένα ε, αυτός είναι ο πιο βασικός κίνδυνος. Μπορούμε να παραμείνουμε βέβαιοι ότι στο μέλλον η πολιτική συνοχή ε, θα τα καταφέρει σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο όπως τα καταφέρνει τώρα ή στο μέλλον ε, υπάρχει ο κίνδυνος πιο κεντροποιημένης πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ. Πρόεδρο ευχαριστώ πολύ. κυρία Νταμάτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους παρισταμένους, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Επίτροπο και τους συναδέλφους. Η δουλειά που μας περιμένει είναι πολύ σημαντική και είναι θεμελιώδης η υπεράσπιση της πολιτικής συνοχής, αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια. Κάτι δεν πάει καλά. Και πλέον υπάρχει ευκαιρία να αλλάξουμε τα πράγματα πρέπει να πούμε ειλικρινώς ότι υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες αναπτύσσονται, αλλά δεν αναπτύσσονται όλες με την ίδια ταχύτητα και νομίζω ότι οι ίδιες είναι αυτές που πάντα υστερούν. Ε, όσον αφορά το ποσοστό της απασχόλησης, μένει χαμηλό και το ποσοστό της ανεργίας είναι υψηλότερο από ό,τι πριν από την κρίση. Οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην παγκοσμιοποίηση, στην ψηφιοποίηση, στην πράσινη ανάπτυξη και στην τεχνολογική αλλαγή. Επομένως δεν μπορούν να ε, προσαρμοστούν στο μέλλον. Και εδώ βλέπουμε κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις ε, και όχι ερωτήσεις. Θεωρούμε καταρχάς ότι το ποσοστό το οποίο προορίζεται για τη μόνη πραγματική ε, συνοχή για την ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει ίδια. Εκφράζουμε τη στεναρή αντίθεσή μας σε ένα μοντέλο οικονομικής διαχείρισης, άμεσης διαχείρισης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα χρηματοδοτεί μόνο προγράμματα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση που σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε τη διαδικασία της εδαφικής συνοχής, δηλαδή έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να συνεχίσετε να χρηματοδοτείτε τις υποδομές μέσω ενισχύσεων και όχι μόνο χρηματοδοτικών μέσων, ακόμα και αν είναι χαμηλού κινδύνου. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αρχιτεκτονική δομή που έχουμε με συνδιαχείριση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κράτη-μέλη και η διαχείριση θα ε, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και των περιφερειών. Ιδιαίτερη προσοχή τώρα στις αρχές διαχείρισης. Γιατί να μην προτείνουμε και να υποχρεώσουμε ε, τη δημοσίευση ενός προγράμματος εργασίας. Δηλαδή, ένα έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι ημερομηνίε για τους διαγωνισμούς για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ώστε να προγραμματίζουμε γέρος ε, και οι επιχειρήσεις αλλά και οι τοπικές αρχές ε, τον τρόπο διαχείρισης. Οι δείκτες. Αναφερόμαστε πάντα στο ΑΕΠ και καλούμε όλους τους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, συμπεριλάβει και άλλους δείκτες πέραν του ΑΕΠ. Παραδείγματος χάρη τον ε, ε, δείκτη κοινωνικής προόδου, αλλά και τον δείκτη καλύτερης ζωής, τον Better Life Index. θεωρούμε ότι τα μέτρα τα οποία συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ταμείων με την υγιή οικονομική διαχείριση και τις κυρώσεις που προβλέπονται, ου μόνο ανακατάλληλες αλλά και αντιπαραγωγικές η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έλεγε στην προηγούμενη έκθεση, στην έκτη έκθεση πρόοδου, ότι οι τοπικές και περιφερειακές ε, αρχές είναι αρμόδιες περίπου για το 30% της κρατικής δημόσιας δαπάνης και περίπου το 60% των κρατικών επενδύσεων. Η αύξηση του δημοσίου χρέους ε, ε, προέρχεται και από τις δραστηριότητες της κεντρικής κυβέρνησης λοιπόν και όχι της περιφερειακής κυβέρνησης ή της τοπικής κυβέρνησης και υπάρχει και θέμα προγραμματισμού και συνδυασμού με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το άρθρο 23 ευτυχώ δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Επομένω πρέπει να περάσουμε στη ρίζα του προβλήματο και να μην ε, κοροϊδευόμαστε με επενδύσει που τελικά οδηγούν στο 0%. Να δούμε το πραγματικό ποσοστό σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και Πολιτική συνοχή διαγράφοντα οποιαδήποτε πρόβληψη για άδικε ε, ε και ιδιαίτερα επαχθεί κυρώσει για τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ και του δικαιούχου των έργων. Η πολιτική συνοχής δεν είναι η αιτία του χρέους. Κάθε άλλο είναι τμήμα μιας πολιτικής ε, επενδύσεων και αν είναι και καλή ε, τότε μπορεί να είναι και μέρος της λύσης. Προτείνουμε λοιπόν αναθεώρηση τη ρήτρα των επενδύσεων ώστε οι περιφερειακές επενδύσεις και οι εθνικές επενδύσεις που θα συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία να εξαιρούνται από τον υπολογισμό των εθνικών ε, ελλημάτων. Τώρα, εμείς ε, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί ένα στοιχείο ευελιξίας ε, το οποίο θα επιτρέπει ε, τη συνδυασμό διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου ε, Στρατηγικών Επενδύσεων. Θέλουμε να έχουμε άμεσες επενδύσεις, όπως για παράδειγμα ε, το Sign of Excellence, το οποίο εγγυάται ότι ε, έχουμε κάποια προγράμματα στον ορίζοντα 2020, τα οποία είναι αναγνωρισμένα. Είναι υψηλή ποιότητα και μπορούν να έχουν ένα πιστοποιητικό αριστεία και επομένω να υπάρχει χρηματοδότηση μέσω των ε, ταμείων αυτών. Μεταρρυθμίσεις ε, διαρθρωτικές και τεχνική συνδρομή. Ε, κάνουμε διάκριση γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία άμεση σχέση της πολιτικής συνοχής με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όπως ε, υποδεικνύεται στις συστάσεις αναχώρα τεχνική συνδρομή και βελτίωση διοικητική ικανότητα ε, συμφωνούμε απολύτω. Είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Και ίσω ε, και είναι και η ανικανότητα τη διοίκηση να συμμετέχει και να προγραμματίζει ε, είναι ε, αιτία της ε, λοιπούς εφαρμογής της πολιτικής συνοχής επιτόπου. Τώρα, οι διαχειριστικές αρχές και οι ελεγκτικές αρχές πρέπει να ελέγχονται καταλήλων. Θα πρέπει να υπάρχει περιτροπή αλλαγή του προσωπικού, να ελέγχεται το θέμα της έγκρουσης συμφερόντων και προτείνουμε ένα ενιαίο αρμόδιο φορέα ελέγχου σε εθνικό επίπεδο που δεν θα έχει καμία σχέση με περιφερειακές και ε, εθνικές αρχές διαχείρισης των κονδυλίων. Ε, τέλος, για να υπάρχει σεβασμός ε, στην ορθή και ομογενή εφαρμογή των κανόνων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτείνουμε να υπάρχουν Ευρωπαίοι ελεγκτές. Ολοκληρώνω για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα των χρηματοδοτικών μέσων και των τραπεζών. Το ποσοστό χρήσης χρηματοδοτικών μέσων θα επεκταθεί πολύ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βάσει όμως των στοιχείων που έχουμε από τους ίδιους τους ε, δικαιούχους και από το ελεγκτικό συνέδριο πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει καλύτερη διαχείριση και θα πρέπει να προτιμούμε ε, τις τράπεζες στις περιπτωσότερες περιπτώσεις. Πρέπει να προσέξουμε και την ε, επιλογή των διαμεσολαβητών ε, με βάση αυστηρά ε, κριτήρια επιλογής, να υπάρχουν τα καλύτερα πρότυπα διαφάνειας και ευθύνης και οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης μέσω διαμεσολαβητών ή τραπεζών που δρούν ως διαμεσολαβητών θα πρέπει να, να συνοδεύεται και από δημοσίευση των πληροφοριών και των λογιστικών στοιχείων αναχώρα το κόστος, η προμήθεια που παίρνουν οι τράπεζες και οι διαμεσολαβητές ε, είναι πολύ ε, υψηλά. Εάν ένα έργο δίνει 100 στο δικαιούχο, πόσο είναι το κόστος ε, της προμήθειας και πόσα από αυτά τα 100 φτάνουν τελικά ε, πραγματικά στο δικαιούχο. Η επιλογή του μέσου, και με αυτό πραγματικά ολοκληρώνω, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο τρόπο και να γίνεται με βάση τον ε, παράγοντα κινδύνου. Προσοχή λοιπόν στα καταπιστευματικά ταμεία, σε άλλες μορφές ομολόγων, και ε, διότι ελοχεύει ο κίνδυνο να έχουμε μία ακόμα φούσκα. Πρέπει να διασώσουμε την πολιτική συνοχή στην οποία εμείς πιστεύουμε ακράδαντα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σπυρίδων. Πρόεδρε, βέβαια το να ε, επιχειρηματολογήσω υπέρ της πολιτικής συνοχής στο χώρο αυτό είναι σαν να κομίζω γκαλάφικα της Αθήνας, όπως λέμε στην Ελλάδα. Αλλά Πρέπει να συγχαρώ όμως την πολύ συστηματική και σημαντική συνεργασία μεταξύ των Προέδρων Ρέντς και Κοτέρ, αλλά και κυρίως και βεβαίως και της κυρίας Επιτρόπου, η οποία ακούραστα έχει μια ουσιαστική παρουσία όχι μόνο σε συνεδριάσεις σαν και αυτές, αλλά και σε κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν το κάνω για φιλοφρόνηση. Θα εστιαστώ μόνο σε ένα συγκεκριμένο θέμα για να αποφύγω τι επαναλήψει των αξιόλογων ομιλητών που μίλησαν προηγουμένω. Και έχοντα μια εμπειρία 20 ετών ω δήμαρχο και ω επικεφαλή περιφέρεια, θα εστιαστώ στην απόδοση, στη βέλτιστη απόδοση των διαχρονικών ταμείων και στην προσθέμενη αξία που αυτά παράγουν σε κάθε χώρα. Και θέλω να πω το εξή. Πολύ φοβάμαι ότι σε κάποιε χώρε, μπορεί αυτό να μην συμβαίνει σε όλε, γιατί έχουμε διαφορετικά συστήματα τοπικών αρχών από χώρα σε χώρα με διαφορετικέ αμοδιότητες και διαφορετικές δυνατότητες η κάθε πόλη, η κάθε περιφέρεια. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές χώρες όπου ο τρόπος που γίνεται ε, η επιλογή του ποιο θα πάρει ένα συγκεκριμένο έργο δεν ευνοεί την ανάπτυξη, αλλά δυστυχώ γίνεται ένας κατάλογος, μια λίστα έργων. Τι εννοώ δηλαδή. Γίνεται ένα call και λέει έχουμε τόσα χρήματα για οδοποιία. Όταν λοιπόν ένας μεγάλος δήμος ή μια περιφέρεια έχει τη δυνατότητα, θα κάνει αυτό το έργο. Και μπορεί τα έργα αυτά να μην υπακούν σε, μια συνολικό, σε ένα συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης, άρα έχουμε σαν αποτέλεσμα και υπό την πίεση της απορρόφησης να έχουμε μια πολύ ωραία λίστα έργων, αλλά μην έχουμε προστιθέμενη αξία που θα προέκυπτε από ένα συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και τη συμμετοχή στις πολιτικές συνοχίες των κρατών εθνών για παράδειγμα θα μπορούσαν τα κράτη-έθνη προκειμένου να μετριάσουν αυτό να εστιάσουν τις πολιτικές τους ώστε να υπάρχουν οι βασικές υποδομές σε μια περιφέρεια ή σε έναν Δήμο για να μπορέσουν π.χ. να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά από τα διαφορετικά ταμεία χρήματα για αναπλάσεις. Θα πρέπει να να είναι υποχρεωμένε να φροντίσουν για τη συντήρηση των ήδη υπαρχόντων έργων που έγιναν από διαφορετικά ταμεία για να μπορούν να αξιοποιήσουν τα επόμενα. Ή θα πρέπει ίσω να φροντίσουν για την ενδοπεριφερειακή συνοχή. Γιατί υπάρχουν αρκετέ περιφέρειες που δεν υπάρχει συνοχή εντό του, και αυτό οφείλεται κυρίω σε ότι ως μοναδικό γνώμονα για τη χρηματοδότηση έχουμε το ΑΕΠ. Και ε, βέβαια δεν σημαίνει τίποτα αυτό, διότι μπορεί μια πόλη ή στην περιοχή μου ένα νησί να είναι αρκετά εύπορο και προηγμένο σε οικονομικά και μέσα στην περιφέρεια να υπάρχουν περιοχές που είναι από τις πιο ε, ιστερούσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πέντε ακόμη ομιλητές έχω στον καταλογό μου. Έχει περάσει όμως η ώρα. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους, αλλά πρέπει να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Οι συντονιστέ μίλησαν εκ μέρου ε, των πολιτικών ομάδων, λέει η πρόεδρο. Θα σα δώσω το λόγο, κυρία Μπρέσο, και θα ήθελα να σα ζητήσω να είστε πολύ σύντομοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. σε κάποιες περιπτώσεις ε, θα πρέπει να γίνεται καλύτερος ο έλεγχος του χρόνου παρέμβασης. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήσεις πολύ σύντομα. Καταρχάς να υπενθυμίσω ότι οι Επιτροπέ ε, Περιφέρειες Ανταγωνιστικότητες υπέστησαν και αυτές μια σοβαρή κρίση ε, στη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης και επομένως η περιφερειακή πολιτική πρέπει να παραμείνει για όλες τις περιφέρειες. Δεύτερον, μια έκκληση στην Επίτροπο Κρέτσου, την οποία ευχαριστώ για την σημερινή της παρουσία. Το θέμα της απλοποίησης είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Ε, γιατί λοιπόν να μην ε, ξεκινήσουμε μαζί με τους αδέλφους από την Επιτροπή των Περιφερειών που με μεγάλη χαρά βλέπω εδώ μια επαλήθευση της έκθεσης που κάνατε. Να ακούσουμε τους χρήστες, αυτούς που χρησιμοποιούν τα κονδύλια και να μας πούνε εάν οι προτάσεις οι οποίες ε, γίνονται για την απλοποίηση είναι καλές ή αν έχουν κάποια καλύτερη να μας κάνουν. Δεύτερον, ε, τρίτον, συγγνώμη, ε, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε την πολιτική συνοχής για όλα. Θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη διάκριση ε, η διαχείριση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και οι πιθανές κυρώσεις για όσους ε, δεν σέβονται το εξάμεινο ε, είναι τελείως διαφορετική από την περιφερειακή πολιτική που έχει τους δικούς τους όρους και τα δικά της στοιχεία επαλήθευσης. Υπάρχουν μέσα και μπορούμε να το επεξεργαστούμε αυτό. Μια τέταρτη πρόταση το Εράσμους των Ερετών. Εγώ ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει ούτε να τα ακούσει, αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αν θέλουμε να βελτιωθεί η ποιότητα της πολιτικής ε, των περιφερειών, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στη γραφειοκρατία, πρέπει να στοχεύουμε και στην ποιότητα του πολιτικού προσωπικού, στη δυνατότητα να αντιληφθεί τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα ε, πρόγραμμα το οποίο είχε δώσει καλά αποτελέσματα και θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και στην πολιτική συνοχή με τη δυνατότητα ανταλλαγών μεταξύ ερετών από διάφορες περιφέρειες στις οποίες πηγαίνουν τα πράγματα καλά και ίσως και από περιφέρειες στις οποίες τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Τελευταίο, διότι επειδή οι στόχοι τη επόμενη προγραμματική περίοδου αρχίζουν να διαφαίνονται σαφώ, γιατί να μην χρησιμοποιηθεί ένα ποσοστό των ε, πόρων που έχουν απομείνει από αυτή την προγραμματική περίοδο για να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Διότι ένας από τους λόγους των καθυστερήσεων είναι το γεγονός ότι οι περιφέρειες μπορούν να αρχίσουν να σχεδιάζουν μόνο όταν έχει κλείσει το πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένα, έχουν λάβει τα κονδύλια και έχει γίνει η κατανομή. Γιατί να μην βοηθήσουμε να προγραμματίσουν ήδη τουλάχιστον σε γενικές γραμμές το μέλλον τους, να ε, ξεκινήσουμε την δημιουργία προγραμμάτων για θέματα τα οποία γνωρίζουμε ότι σίγουρα θα υπάρχουν. Για παράδειγμα, ενεργειακή πολιτική, η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών την ανταγωνιστικότητα και το ψηφιακό θεματολόγιο. Έτσι θα είναι έτοιμοι και όταν ε, ε, φτάσουν τα κονδύλια θα ξεκινήσει και ο προγραμματισμός. Ο κύριος Κατσιφάρας για πέντε λεπτά παρακαλώ. Δύο λεπτά, συγγνώμη. Νομίζω ότι η συζήτηση γίνεται σε πολύ κρίσιμη χρονική περίοδο για την ίδια την πολιτική συνοχή. Πρέπει όμως να δώσουμε σαφείς απαντήσεις ή να αναζητήσουμε απαντήσεις. Πρωτίστως πολιτικές. Η πολιτική συνοχής ήρθε να δώσει μια απάντηση στην άρση των ανισοτήτων και ταυτόχρονα να διαμορφώσει ένα πλαίσιο ίσων ευκαιριών τέσσερα, τέσσερες περίοδοι με κεντρικό πυρήνα την άρση των ανισοτήτων σήμερα ένας απολογισμός για κάποιες χώρες δεν είναι καλός. Οι ανισότητες έχουν διευρυθεί, οι θέσεις εργασίας που έχουν παραχθεί ή όποιες θέσεις είναι χαμηλού, χαμηλής οικονομικής αμοιβή, είναι πιο φτωχότεροι οι άνθρωποι και η νεολαία σε μεγαλύτερο αδιέξοδο. Άρα λοιπόν είναι η κρίσιμη ώρα να πάρουμε τις σοβαρές αποφάσεις. Η συνοχή θα επηρεάσει και τον πυρήνα της Ευρώπης ως οντότητα. Όχι γεωγραφική απλά, αλλά ως μια οντότητα αξιών, πάνω στην οποία έχει χτίσει την αλληλεγγύη, την παιδεία, την κουλτούρα, την ειρήνη. Άρα λοιπόν θέλουμε πολιτική συνοχής. Ναι, το πλαίσιο που έβαλε η Επίτροπος με τους τέσσερους πυλώνας είναι μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Βεβαίως. Και θα έλεγα περισσότερο ο πρώτος πυλώνας που είναι η εμπιστοσύνη. Το πολιτικό πρόβλημα της Ευρώπης είναι το τεκμήριο εμπιστοσύνης έχει χαθεί από τις τοπικές κοινωνίες. Εδώ αν θέλουμε να χτίσουμε μια άλλη Ευρώπη με ελπίδα, με συμμετοχή, πρέπει να πατήσουμε πάνω σε αυτό τον πυλώνα. Υπάρχουν οικονομικά εργαλεία που δεν φτάνουν στις χώρες μας. Τελειώνω. Π.χ. το πακέτο Γιούγκερ. Δεν είναι θέμα μόνο μια αδυναμίας. Είναι θέμα το μοντέλο παραγωγής που έχουμε. Δεν απαντά. Άρα εκεί πρέπει να απαντήσουμε. Θέλω να τελειώσω ότι θέλουμε την πολιτική συνοχής, πρέπει να ξαναδούμε τα σημεία εχμής, νεολαία, φτώχεια, περιφέρειες σε κίνδυνο και να συγχαρώ και δημόσια την κυρία Επίτροπο, την κυρία Κρέτσου. Έχει δώσει δείγματα γραφής και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τουλάχιστον στη χώρα μου. Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι και σε άλλες χώρες. Δεν είναι μόνο η φυσική της παρουσία εκεί. Είναι η ποιότητα της πολιτικής και των προτεραιοτήτων που θέτει. Ε, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα κέρδος και για την Ευρώπη. Το λέω δημόσια, σπάνια μας δίνεται αυτή η δυνατότητα και νομίζω ότι με τους πυλώνες που θέσατε πρέπει να ταρακουνήσετε και λίγο παραπάνω την Ευρώπη. Κυρία Κρέτσου, μην διστάσετε. Ταρακουνήστε την παραπάνω. Γιατί η συνοχή θα δώσει απάντηση στο πολιτικό διακύβημα της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μπόκοβιτς, παρακαλώ πολύ σύντομα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η πολιτική συνοχή είναι μία από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά το γεγονός ότι αποτελεί μόνο το 0,3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στις εθνικές πολιτικές ε, μέσω διαφόρων ε, ε, διάβλων. Ο συνάδελφος από την Ιρλανδία μας μίλησε για την κατάσταση εκεί, τώρα και στο παρελθόν. Ο, επίσης, ε, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πραγματικά διευκολύνθηκε πάρα πολύ από την πολιτική συνοχή. Ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια στα νέα κράτη-μέλη. Έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και Κατά τα τελευταία χρόνια έχουμε όλο και, περισσότερο, όλο και περισσότερη δυσκολία ε, να δείξουμε τα αποτελέσματα της ε, συνοχής ε, στους πολίτες μας από την περίοδο, την περίοδο 2012 έως 2016 έχουμε πάρα πολλές επενδύσεις ε, ε, και στη, στην, ε, σελίδα 178 της, της έκθεσης για την πολιτική συνοχή φαίνεται αυτό, φαίνεται δηλαδή ότι υπήρξαν προβλήματα με ε, την ε, διανομή των πόρων. Πρέπει αυτό να διορθωθεί στο μέλλον. δεν ε, υπάρχουν μετανάστες σε όλες τις περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των πόλεων και των περιοχών της υπαίθρου. αυξήθηκε κατά 12% σε μερικές περιφέρειες από το 2012 στο 2016 ανεργία. Σε άλλες ε, περιφέρειες όμως ήταν ε, πιο ε, σταθερή η κατάσταση. Εγώ συμμετέχω σε μεγάλο βαθμό στο εγχείρημα των εφιών πόλεων. Πρέπει να υπάρξουν νέε θέσει απασχόληση και καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ε, πρέπει να υπάρξει μια ευφυής ρύθμιση. Οι προκλήσεις που υπάρχουν στις πράσινες θέσεις απασχόλησης, ε, στην ε, ενεργειακή ένωση, τα ζητήματα της ενέργειας, όλα αυτά είναι ευκολότερο να τα αντιμετωπίσουμε μέσω της πολιτικής συνοχής και χαιρόμαστε όλος ιδιαιτέρως που μεταξύ ημών βρίσκονται άνθρωποι που δουλεύουν για, αυτές, ε, για, αυτά, για αυτούς τους στόχους στις περιφέρειες γιατί εκεί θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην πολιτική συνοχή. Thank you very much. I would like... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να καλωσορίσω την έκθεση για τη συνοχή γιατί επικεντρώνεται στην ε, αποτελεσματικότητα βάσει των επιτευγμάτων που έχουν ε, σημειωθεί σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δύο ερωτήσει ε, ανακύπτουν ε, από την έκθεση. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση της εφαρμογής στην τρέχουσα περίοδο και κατά δεύτερον, πώς θα προετοιμαστούμε καλύτερα για την μελλοντική περίοδο πώς θα σημειώσουμε πιο μεγάλη επιτυχία και σε ό,τι αφορά και τη διαδικασία σύγκληση. Αν θέλουμε λοιπόν να απαντήσουμε στα δύο ερωτήματα, καταρχάς για το πώς θα επιταχυνθεί η υλοποίηση και η εφαρμογή, φυσικά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι λείπουν και δεν υπάρχουν επαρκή προγρήματα, ε, ότι υπάρχουν ελλείμματα στις υποδομές και στις ε, δυνάμεις μας ε, και η απάντηση σε όλα αυτά είναι μία μόνο. Διευθυντικές μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά χωρίς μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, στο δικαστικό σώμα, στις επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Φυσικά λοιπόν αυτά θα πρέπει να γίνουν τώρα προκειμένου να έχουμε επιτυχία στο μέλλον γιατί δεν μπορούν να επιληθούν όλα αυτά γρήγορα και να υπάρξει επιτυχία και τα αποτελέσματα που θέλουμε στην τρέχουσα περίοδο. Αλλά ενδεχομένω μπορούμε να δούμε τι μέτρα χρειάζονται στην τρέχουσα περίοδο. Για παράδειγμα, μιλήσατε για την αλλαγή των κανονισμών σε ό,τι αφορά τις φυσικές καταστροφές. Πάρα πολύ θετικό και αυτό. Γιατί προσπαθούμε με κάποιο τρόπο με την πολιτική συνοχή να δώσουμε μία απάντηση στι ανάγκες, στις πρακτικές ανάγκες των πολιτών. Να υποστηρίξουμε τι χρειάζεται δεν χρειάζονται στην πράξη. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και άλλα μέτρα. Για παράδειγμα, για την περίοδο 2007-2013 εισαγάγατε την ευελιξία μεταξύ των προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τα προγράμματα για να υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθούν πόροι από τομείς με πλεόνασμα σε τομείς με έλλειμμα. Θα πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε με συγκεκριμένα μέτρα και μέσα για συγκεκριμένα προβλήματα, για συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Και στην τελική ανάλυση, όταν σκεφτόμαστε το μέλλον, θα πρέπει να δούμε τι χρειαζόμαστε για να πετύχουμε υψηλότερο ποσοστό επιτυχία σε περιοχές που μένουν πίσω. Και φυσικά ένα καλό μείγμα οικονομικής πολιτικής. Δεν μπορούμε να επιδροθούμε μόνο στις επενδύσεις, θα πρέπει να κοιτάξουμε και τις δρατικές μεταρρυθμίσεις, το οποίο και το υπογραμμίσατε και επίσης έξυπνη δημοσιονομική ενίσχυση. Θα πρέπει προς το σκοπό αυτό να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία με τους εθνικούς προϋπολογισμούς και επιτροπέ μιλήσατε για νέες προτεραιότητες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην πολιτική συνοχή. Αλλά πίστευω ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο περιθώριο για νέες προτεραιότητες και αυτό γιατί η πολιτική συνοχή είναι περιορισμένη λόγω του ευρωπαϊκού προπολογισμού που είναι περιορισμένος αλλά χρειάζονται ακριβώς μια συνέργεια με τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Γιατί έτσι από κοινού ενδεχομένω κάτι παραπάνω να πετύχουμε και σε ό,τι αφορά επίση τι διαθετικέ μεταρρυθμίσει, χρειαζόμαστε πιο πολλέ δράσει από του εθνικού προπολογισμού σε εθνικό επίπεδο, αλλά επίση μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και των λειτουργικών προγραμμάτων, γιατί τα εθνικά προγράμματα είναι για τρία η τριετή περίοδο, ενώ τα λειτουργικά προγράμματα έχουν επταετή περίοδο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συνεργία μεταξύ αυτών. Ευχαριστώ κύριε Νίλσεν, έχει το λόγο. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, Χαίρομαι πολύ που βλέπω την άποψή σας για το ενιαίο σύνολο κανόνων ε, για ε, τα κονδύλια στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, αλλά γνωρίζουμε ότι η γραφειοκρατία που συνδέεται ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προγράμματα της δημιουργείται στα κράτη-μέλη για τον τρόπο, από το, λόγω του τρόπου με τον οποίο έχουν δομηθεί οι διοικητικέ υπηρεσίες εκεί. Οπότε το ερώτημά μου είναι αν τα κράτη-μέλη θα δεχθούν ε, ένα σύνολο κανόνων ε, το οποίο θα επιφέρει ακόμη περισσότερη γραφειοκρατία ή αν θα είστε πιο αυστηρίως προς αυτό. Να δώσω τώρα το λόγο στην Επίτροπο να απαντήσει στις ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Μερικές ερωτήσεις δεν ήταν και πολύ εύκολες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τι τόσο ε, καλές ε, ιδέες. Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχο της σημερινής ε, συνεδρίασης, να σας ακούσω. Οπότε, όπως είπα, για να απαντήσω στην κριτική ότι δεν είμαστε πολύ συγκεκριμένοι με τις προτάσεις μας, Κοιτάξτε, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει το Μάιο του 2018 την πρότασή της για τον προϋπολογισμό και έχει αρχίσει τώρα αυτή η συζήτηση και στο τέλος του έτους ε, θα ξεκινήσει μια ευρεία δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και βεβαίως ε, σας ενθαρρύνω όλους ε, να ε, συμμετάσχετε και από την Επιτροπή Κοτέρ και από την Επιτροπή Ρέτζι. Είστε οι πιο σημαντικοί μας εταίροι γιατί έχετε τόσες πολλές ιδέες, εσείς ε, εργάζεστε επί των, ζητημάτων αυτών. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις, δεν νομίζω ότι θα καταφέρω να απαντήσω σε όλες, αλλά θα προσπαθήσω κάπως να ομαδοποιήσω τις απαντήσεις μου αυτό που είπε ο κύριος Φανίστελρο θα το πάρω ως ε, σύνθημα ότι πρέπει να δράσουμε και όχι να περιμένουμε. Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι το σύνθημά μας ε, για, τις, ε, για τους επόμενους μήνες. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για την καθημερινή μας εργασία. Κάθε φορά πριν από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε πολλές συζητήσεις να κάνουμε αυτή τη φορά, όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα κάθε ιδέα από εσά, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Επιτροπή Περιφερειών, είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτες και για να απαντήσω απευθείας ε, στην ιδέα αυτή του εξυγχρονισμού εγώ πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να κάνουμε έναν εξυγχρονισμό όντω και μερικέ φορέ είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και άλλε φορέ πολύ ευέλικτοι με τα κράτη-μέλη. Για τον ΙΣΙΝ 2. Νομίζω ότι ήταν ένα κίνητρο, τότε σκεφτόμασταν ότι επρόκειτο για ένα κίνητρο, αλλά σήμερα διερευνούμε τη δυνατότητα επανεισαγωγής ε, του νησιν ε, 2 γιατί κατά τη γνώμη μου θα συνεισφέρει στην επίσπευση της ε, εφαρμογής αν βέβαια συνδεθεί με περισσότερα στρατηγικά προγράμματα. Οπότε κύριε Φανίστελ, δίκιο έχετε ε, ότι ε, το ΣΕΦ δούλευε γιατί υπήρχε μια, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μεταξύ μας όλα τα προγράμματα που ήταν έτοιμα υπό τη δική μας πολιτική συνοχή για τις μεταφορές, τα κράτη-μέλη τα ενέτασαν στο ΣΕΦ γιατί θεωρούσαν ότι θα είχαν χρόνο μέχρι το 2023 και σε πολλά κράτη-μέλη είμαστε τώρα σε μια κατάσταση ε, στην οποία δεν υπάρχουν νέα προγράμματα υποδομής για τις μεταφορές, γιατί ό,τι έχουν ε, το εντάσσουν στο ΣΕΦ για να μπορούν να ξοδέψουν τα χρήματα στην προθεσμία των τριών ετών. Οπότε τα κράτη-μέλη, αν ε, υποστούν πίεση, θα ε, επιφέρουν αποτελέσματα. Αν όχι, καθυστερούν αν είμαστε ευέλικτοι. Γι' αυτό υπάρχει τόσο χαμηλός ρυθμός υλοποίησης αρχίζουν αλλά έχουν τις προκαταβολές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, έχουν τώρα χρόνο μέχρι το 2020, μετά μέχρι το 2023, οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι είναι προς το συμφέρον των πολιτών, γιατί εμείς δουλεύουμε πολύ σκληρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο ΚΟΤΕΡ, στην Ευρωπαϊκή, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ε, Επιτροπή Ρέτζι, όμως έχουμε υπάρχει αρκετό, υπάρχουν αρκετά αποτελέσματα. Νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε λοιπόν τον ΙΣΙΝ 3 ξανά. Πολύ προσεκτικά κύριε Όσβαλντ. Ε, εμείς παρακολουθούμε τις ε, γνωμοδοτήσεις της ΚΟΤΕΡ ε, με πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε πάρα πολλές ανισότητες μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης και μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Πράγματι πρέπει όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για αυτήν την πρωτοβουλία για τις ε, περιφέρειες που καθυστερούν, ε, γιατί υπήρξαν πολλές ερωτήσεις από εσά, από τον κύριο Ποτολίν, από την κυρία Νταμάτο. Ε, υπάρχουν λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες που καθυστερούν. Έχουμε μια πρωτοβουλία για αυτές και θέλουμε να τις βοηθήσουμε. Πρέπει να είμαστε σαφείς ότι η έκθεση αυτή δείχνει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ε, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φοβάται ε, την αλλαγή. Ε, οι περιφέρειες αυτές έχουν, ε, παρουσιάζουν μειωμένη ε, βιομηχανική δραστηριότητα, χάνονται θέσεις εργασίας, μειώνονται οι μισθοί και υπάρχει πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση και για τους υπαλλήλους είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενθουσιασμός για την αξιοποίηση των κονδυλίων, για την ανάληψη νέων πρωτοβουλειών ε, και όλα αυτά στις περιοχές που καθυστερούν και που αντιμετωπίζουν προβλήματα ε, είναι πολύ περιορισμένο. Ο ενθουσιασμός αυτός είναι πολύ περιορισμένος. Έχουμε επίσης ε, να ασχοληθούμε και με τα ε, συναισθήματα, να λάβουμε υπόψη ε, και την ε, συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων επιτόπου. Αλλά η εδαφική συνοχή που είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε και από τον κύριο Ζάγκρα, από τον κύριο Κοτσολίνο, από την κυρία Νταμάτο και από άλλα μέλη των επιτροπών νομίζω ότι ε, πρέπει να προσεχθούν περισσότερο. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια πιλωτικά προγράμματα για να ε, συνοδεύονται ήδη από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο κάποιες ε, περιφέρειες οι οποίες δεν τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά με όλες αυτές τις αλλαγές και εμείς θα είμαστε και παρόντες επιτόπου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις περιφέρειες αυτές να υποστηρίξουν ε, τις περιφέρειες αυτές τη βιομηχανική μετάβαση και την οικονομική τους ε, ε, εξέλιξη. Εμείς συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορούμε να βοηθήσουμε στην ψηφιοποίηση και την ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων. Ε, πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση της πολιτικής αυτής κατά τη γνώμη μας και πρέπει να εστιάζουμε περισσότερο στους ε, κινητήριους μοχλούς ε, της ανάπτυξης που είναι βεβαίως η καινοτομία και η εκπαίδευση και η διοικητική ικανότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως είπα λοιπόν κύριε Κοτσολίνο εγώ ανησυχώ όλους ιδιαίτερος για όλες αυτές τις περιφέρειες που καθυστερούν, που υπάρχει μείωση της ανάπτυξης συνεχώς και εσείς και η κυρία Νταμάτο προέρχεστε από μία περιοχή στην οποία επενδύουμε τόσα πολλά χρόνια χωρίς ε, να υπάρχει η απαραίτητη ανάπτυξη ε, και υπάρχει μάλιστα και έλλειψη ανάπτυξης παρά το γεγονός ότι εδώ και δεκαετίες επενδύουμε. Είναι λοιπόν ε, σημαντικό να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα για τις περιφέρειες αυτές ε, γιατί υπάρχουν περιφέρειες που ξεκινούν από την αρχή, αλλά όταν υπάρχουν επενδύσεις ε, υπάρχουν και αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως και άλλες περιφέρειες όπου δεν υπάρχουν αποτελέσματα και αυτό ε, πρέπει να συνδέεται με διαρθρωτικές αλλαγές, γιατί αυτές οι επενδύσεις, κατά την εμπειρία μας, σύμφωνα με την εμπειρία μας, ε, δεν έχουν αποτέλεσμα αν γίνονται μεμονωμένα. Πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση με την, της πολιτικής συνοχής με την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης. Αυτό είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα δαπανώνται αποτελεσματικά. Και βεβαίως ε, σας ε, διαβεβαιώ ότι θα είναι αναλογική ε, και θα παρέχει τα σωστά κίνητρα αυτή η προσέγγιση. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαμε να το δούμε και αντιστρόφως, όχι ως τιμωρία, αλλά ως θετικό κίνητρο για τα κράτη-μέλη, να υπάρχει μια επιβράβευση για τις ε, επιτυχημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τους, ε, οπότε κατά τη γνώμη μου οι κυρώσεις δεν λειτουργούν Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με όλα τα κράτη-μέλη για να αποφύγουμε την αναστολή ε, των κονδυλίων. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει αναστολή πληρωμών για αυτή την προγραμματική περίοδο καθόλου. Οπότε, όπως είπα, για τις ε, περιφέρειες ε, που καθυστερούν, εγώ είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σας επί του θέματος αυτού, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό Έχουμε και εμείς τις δικές μας μελέτες και έχουμε διαπιστώσει ότι αυτές οι περιφέρειες έχουν χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλό ε, ποσοστό απασχολησιμότητας. Αυτός ο, αυτή η έλλειψη επιχειρηματικού δυναμισμού έχει να κάνει και με το σύστημα καινοτομία όλων αυτών των ε, περιφερειών. Γι' αυτό θέλουμε να υποστηρίξουμε την πρότασή σας ε, για την ευφυή εξειδίκευση, η στρατηγική με την οποία βασιζόμαστε τα ισχυρά σημεία αυτών των περιφερειών. Δεν μπορούμε να έχουμε 300 περιφέρειες στην Ευρώπη που να μοιάζουν με την κοιλάδα του πυρητίου, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε αγροτουρισμό, έχουμε την ε, αεροδιαστημική στην, ε, στις κάτω χώρες. Ε, υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε για να στοχεύσουμε την αντιμετώπιση των εμποδίων που έχουμε μπροστά μας. Η θεσμική υποδομή, η δεσμική ικανότητα είναι κάτι άλλο, ε, το οποίο επίσης συνδέεται με περιοχές, περιφέρειες που καθυστερούν ε, ή που παραμένουν ε, σε μια κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα που λιμνάζουν, θέλουμε να αυξήσουμε τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, ε, να υπάρχει εξυγχρονισμός του συστήματος δημοσίων προμηθειών, ενίσχυση ε, της καταπολέμησης της διαφθοράς. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα αυτή της κυρίας Μπρέσο να υπάρχει αυτό το εράσμους για τους ε, εκλεγέντες εκπροσώπους. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε σε υψηλού επίπεδου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι είναι κακή ιδέα καθόλου. Σε πολλά κράτη-μέλη θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ξέρω ότι υπήρξε μια τέτοια απόπειρα στο παρελθόν, αλλά υπήρξε πολύ μεγάλη αντίσταση σε αυτή την ιδέα, γιατί υπάρχει αυτή η ιδέα ε, ότι το Εράσμους αφορά περισσότερο φοιτητές, ε, ανταλλαγή απόψεων... Όμως ε, υπάρχει ε, συνεργασία ομοτήμων ε, στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων μπορούμε να κάνουμε και το ίδιο για τους πολιτικούς, ανταλλαγή απόψεων για βέλτιστες πρακτικές, πώς μπορεί να συμπεριφέρεται κάποιος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τη στιγμή που θα έχει εκλεγεί. Όσον αφορά τώρα το θεματολόγιο για τις πόλεις, ε, εγώ θα ήθελα να προχωρήσω πέρα από αυτό, πέρα από αυτό το θεματολόγιο, αλλά δεν θέλω να χάσω αυτήν την ευκαιρία να αποτίσω φόρο τιμής ε, στο δήμαρχο του Άμστερνταμ, τον οποίο χάσαμε την περασμένη εβδομάδα ήταν πυλώνας για μας, ήταν ένας από εκείνους που μας βοήθησε πάρα πολύ να την εγκρίνουμε και το σύμφωνο του Άμστερνταμ επίση και δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα σε αυτό το σημείο με το θεματολόγιο αυτό χωρίς τον κύριο Βαντερφάν οπότε δεν ξέρω αν τον είχατε γνωρίσει. Νομίζω πάντως ότι από άποψη διοικητικής ικανότητας ε, ήταν πραγματικά ο πιο λαμπρός δήμαρχος που έχω γνωρίσει συνεργάστηκε μαζί μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θεματολόγιο αυτό ε, και θα έρθει στα χέρια σας με μια έκθεση σχετικά είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ε, των δημάρχων ε, με εμά. Θα ήθελα όμω να το αναφέρω αυτό για το δήμαρχο του Άμστερνταμ, γιατί πραγματικά ήταν υποστηρικτή μα εντός τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να έχουμε αυτό το θεματολόγιο, ε, στον αγώνα μας να υπάρξει αυτό το θεματολόγιο, έγραψε μία επιστολή στο, στους πολίτες του Άμστερνταμ όταν έμαθε ότι είχε αρρωστήσει, είχε το σθένος να μιλήσει απευθείας με τους πολίτες, ε, τους είπε να φροντίζουν ο ένας τον άλλον και την πόλη τους και νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για, για πολλούς από εμά. Τώρα για το ερώτημα του Σουηδού συναδέλφου για τους ευάλωτους ανθρώπους, τους ηλικιωμένου. Είναι πολύ σημαντικό για μας και η μετανάστευση φυσικά. Ενθαρρύνουμε όπως γνωρίζετε όλα τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια μας όχι μόνο ε, κατεπηγόντως στην περίπτωση των μεταναστών αλλά και για την ένταξη γιατί χωρίς την ένταξη θα μπορούσε να είναι ατομική βόμβα στο μέλλον η, η για τις μελλοντικέ γενναίες. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε για να υπάρξουν μέτρα άμεσα να ε, υποδεχθούμε τους ανθρώπους αυτούς ε, για τη γλώσσα, για τα σχολεία. Ε, υπάρχει υποδομή των κοινωνικών ταμείων αλλά και το ΆΜΙΦ το οποίο ε, διαχειρίζεται η αρμοδιότητα του κυρίου ε, Αβραμόπουλου. Νομίζω η έγκριση της ε, διασυνοριακής επικοινωνίας ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ήταν νομίζω ένα από τα βασικά επιτεύγματα αυτής της ε, χρονιάς μαζί με το αστικό θεματολόγιο. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μία ε, ανακοίνωση σε σχέση με το θέμα αυτό υπάρχουν ήδη κάποια αποτελέσματα σε σχέση με την περιφερειακή πολιτική του τρέχοντος έτους αυτό το ζήτημα της συγχρηματοδότησης που θέσατε. Κατά τη γνώμη μου, ε, αυτό το υψηλό επίπεδο συγχρηματοδότησης δικαιολογείται σε δύσκολες οικονομικές ε, συνθήκες και πρέπει να κάνουμε μία αξιολόγηση. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ ευχάριστο για τα κράτη-μέλη να το ε, σκέφτονται αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη οικειοποίηση και πιστεύω επίσης ότι πρέπει να επισπευθεί η εφαρμογή. Όσον αφορά τη δική μας την ανακοίνωση, Νομίζω ότι υπήρξε μια ανακοίνωση πέρσι. Εδώ και πολλούς μήνες προσπαθούμε να ε, αυξήσουμε την ορατότητα των πολιτικών μας. Στο Συμβούλιο υπό την Προεδρία της Μάλτας ε, ε, υποβάλαμε 7 ιδέες στα κράτη-μέλη. Η συνάδελφός μου, η κυρία Τάισεν από το Βέλγιο και Είμαι πολύ ευγνώμων στην Επιτροπή Περιφερειών για τη συνεργασία, γιατί νομίζω ότι έχει έρθει επιτέλους ο καιρός, όχι μόνο για μας, αλλά για τους δικαιούχους, ε, ε, τους νομικούς, τους γιατρούς, ε, τους εκπαιδευτικούς, να μιλήσουν για την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Το Ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι 78% όσων έχουν ακούσει τις πολιτική, την πολιτική ε, αυτή έχουν μια πολύ θετική εντύπωση. Το ερώτημα είναι ότι 70% ε, περίπου 30% ε, δεν έχουν καν ακούσει όταν λοιπόν πηγαίνουν στα σχολεία ή στους αυτοκινητοδρόμους δεν σκέφτονται ότι όλα αυτά γίνονται με ευρωπαϊκό χρήμα. Για το ερώτημα τώρα ε, του 20% της πολιτικής συνοχής για την ε, ενεργειακή μετάβαση, ε, το κλίμα. Εμείς με τον Επίτροπο Κανιέτε και με τους Επιτρόπους Κανιέτε και Σεύτσοβιτς το έχουμε συζητήσει και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, για τον πλανήτη μας να πρωτοστατήσουμε ειδικότερα για την COP του 2020 και το πώς καταραίουν οι ε, σχετικές συνομιλίες. Όμως πρέπει να ε, συνεχίσουμε με την ενεργειακή μας μετάβαση και την, την αλλαγή της οικονομίας μας προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τα μεγάλα ποσά ε, που έχουν στη διάθεσή τους για την ενεργειακή αποδοτικότητα, για τους νέους δείκτες. Ήταν μια συζήτηση που μένεται εδώ και τρία χρόνια ε, ξέρω ότι την έχετε κάνει κι εσείς εδώ στην Επιτροπή Ρέτζη. Εντάξει, το κατακεφαλήνα ΕΠ δεν είναι το καλύτερο, ο καλύτερος δείκτης, αλλά τότε υπήρχε συνένεση. Κατά την τελευταία περίοδο βέβαια ε, διαπιστώνουμε και το γνωρίζετε ότι το κατακεφαλήνα ΕΠ δεν είναι μοναδικός δείκτης και δεν μας δίνει τις αποχρώσεις της ε, πραγματικότητας. Εγώ λοιπόν προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει πραγματικά να λάβουμε υπόψη ε, την ιδέα εισαγωγή δικτών που είναι πιο σημαντική για την ποιότητα της ζωής όπως κοινωνική ένταξη, φτώχεια, ανάπτυξη γιατί εδώ είμαστε στο Βέλγιο Έχουμε υψηλό κατακεφαλήν ΑΕΠ, όμως ε, εξακολουθούν ε, να υπάρχουν πολλά ε, τμήματα της περιφέρειας με υψηλά ποσοστά φτώχειας και ενεργείας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβληματιστούμε περισσότερο επ' αυτού. Εμείς θέλουμε να διερευνήσουμε και άλλες εναλλακτικές επιλογές με τον ΩΣΑ, με την Παγκόσμια Τράπεζα και θα θέλαμε να συνεργαστούμε και με εσά για να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τους κατάλληλους δείκτες Όσον αφορά τώρα την ε, καταπολέμηση της ανεργίας, πρέπει να πω ότι όχι μόνο το κοινωνικό ταμείο, αλλά όλα τα διαρθρωτικά ταμεία καταπολεμούν την ε, ανεργία και αυτό είναι ο βασικός μας στόχος. Κύριε Κατανέου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ε, λόγια σας. Είστε πάρα πολύ αισιόδοξο. Λειτουργεί η πολιτική συνοχή, αλλά όπως είπατε υπάρχουν χώρες στις οποίες άνω του 50% των δημοσίων επενδύσεων εξαρτώνται από τα δικά μας τα κονδύλια. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινεί, γιατί μεταξύ μα είμαστε και θεωρούμε ότι υφίσταται επίθεση η συγκεκριμένη πολιτική ε, είπα νέε προκλήσει, όχι νέε προτεραιότητε. Έχουμε πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις ε, για το Brexit, για παράδειγμα. Πώς ε, θα καλύψουμε το κενό. Δεν ξέρουμε πώς ε, θα ληφθούν υπόψη η εσωτερική, εξωτερική ασφάλεια, ο Ευρωπαϊκός στρατός, η μετανάστευση, όλα αυτά. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουν. Η δική μου άποψη λοιπόν είναι ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και πρέπει να έχουμε και ε, τον αντίστοιχο προπολογισμό, να θέλουμε τα ίδια ποσά. Αν δεν είμαστε φιλόδοξοι, αν δεν συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη ώστε να δούμε πώς μπορούμε να ε, επεκτείνουμε τους πόρους μας ε, και ε, να δούμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη να ενδιαφέρονται να καλύψουν το κενό, ενδεχομένως η πολιτική συνοχής να έχει μικρότερη εμβέλεια. Εγώ τουλάχιστον πάντως προσπαθώ σε αυτό το έγγραφο θέσης να αγωνιστώ, να παραμείνει η, πολιτική συνοχής στα ε, ίδια επίπεδα. Νομίζω ότι πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή να καταπολεμήσουμε τις προκαταλήψεις ότι είναι ε, παλιά αυτή η πολιτική συνοχής. Ε, εντάξει, είναι γεγονός ότι δεν έχει μεταρρυθμιστεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως είναι σύγχρονη και μπορούμε να την προσαρμόσουμε στις αναδυόμενες προκλήσεις. Υπήρξε μία ερώτηση για τις εκ των προτέρων ερεσιμότητε, νομίζω ότι έχουν απτά αποτελέσματα οι αιρεσιμότητε αυτές ως προϋπόθεση για, την, ε, για τις επιτυχείς ε, επενδύσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτές ε, τις αιρεσιμότητε στο μέλλον, αλλά πρέπει να τις απλοποιήσουμε και να τις ευθυγραμμίσουμε. Για τις τοπικές αρχές, ναι, έχουν έναν βασικό ρόλο να διαδραματίσουν, γιατί γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση επιτόπου. Χρειαζόμαστε εδώ δηλαδή την επικουρικότητα και την επικουρικότητα. Κύριε Σπυρίδωνα, αναφερθήκατε κι εσείς ε, ε, στο ρόλο των τοπικών ε, αρχών. Ξέρετε ότι υπάρχουν οι συμφωνίες συνεργασίας, υπάρχουν, υπάρχει αυτή η στρατηγική προσέγγιση και οι σχετικές συμφωνίες, ότι υπάρχουν λεπτομερείς δράσεις για να μπορέσουμε να επιτύχουμε στρατηγικούς στόχους. Κυρία Πρέσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλοποίηση ήταν πράγματι η προτεραιότητά μου για τον πρώτο μήνα. Είχαμε αυτό το υψηλό, την ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλοποίηση ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει και ένα από τα μέτρα αυτής της ε, προγραμματικής περίοδου που θα επιζήσει. Επίσης αυτό το omnibus, ε, η διαδικασία omnibus ελπίζω να συνεχιστεί για να μπορούν οι δικαιούχοι να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα μέτρα, να τα αξιοποιήσουν. Πάντως πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ε, θέλουμε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και θα πρέπει να το προωθήσουμε. Κύριε Κατσιφάρα, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά όλα τα κρατημέλη, σας διαβεβαιώ, ε, είναι ε, στην καρδιά, στο επίκεντρο των επιχειρησιακών πολιτικών μας. Ε, ξέρουμε ότι υπήρχε μια έκτακτη κατάσταση κατεπίγουσα στην Ελλάδα. Ήμασταν εκεί, ήμασταν εκεί και όταν χρειάστηκε και στην Ιταλία. Ε, προσπαθούμε ε, να βοηθήσουμε και στην περίπτωση της Ελλάδας αλλά και στην περίπτωση των θεομηνιών όχι μόνο για την Ιταλία αλλά και άλλες χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 95% για την ανοικοδόμηση οπότε πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, το είπα αυτό για να μην υπάρχουν αυτές οι μακροχρόνιες διαδικασίες ε, με κρίσεις απρόβλεπτες. Όσον αφορά την εφαρμογή, ε, αναφερθήκατε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, έχει φύγει, δεν εδώ. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν ε, ανομαλίες, αλλά μπορώ να το πω για όλους ότι η εφαρμογή επιτόπου επιταχύνεται για αυτή την προγραμματική περίοδο, έχει βελτιωθεί η επιλογή των ε, έργων, έχει φτάσει στο 40% ε, της πολιτικής συνοχής και 24% των ε, βασικών προγραμμάτων έχουν ήδη κατατεθεί για να εγκριθούν. Οπότε πρέπει να πω ότι συνεχίζει η επίσπευση ε, για την υλοποίηση, την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τώρα προσπαθούμε να δούμε τα προγράμματα που προχωρούν αργά για να δούμε πώς με τις τοπικές αρχές μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Για το τελευταίο ερώτημα του κυρίου Νίλσεν, ξέρετε ότι εγώ είμαι πολύ ανοιχτή ε, για να απομακρύνουμε όλους ε, τους ε, άχρηστους κανόνες, 600 σελίδες κανονισμού, 2.000 σελίδες ε, κατευθυντήριες γραμμές γιατί δεν ήξεραν πώς να ερμηνεύσουν το κανονισμό το δικό σας, ε, του ε, Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ε, έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να κάνουμε, πρέπει πάντως να είμαστε βέβαιοι για τις συνέπειες και πρέπει να είμαστε σκληροί με τα κράτη-μέλη γιατί προσθέτουν, προσθέτουν, προσθέτουν για να καλύπτονται. Όταν όμως βλέπει κανείς τι γίνεται επί τόπου, ο κόσμος λέει «Α, δεν θέλουμε, ευχαριστούμε πολύ, δεν θα πάρουμε άλλα από αυτά τα διαρθρωτικά ταμεία γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκα». Δεν είμαι υπέρ ε, λοιπόν όλης αυτής της κατάστασης. Στον ε, 21ο αιώνα ζούμε. Δεν θεωρώ λογικό να υπάρχουν ε, τώρα έργα, ε, προγράμματα με 700 σελίδες. Όλα τα κράτη-μέλη θέλουμε και ζητούμε ηλεκτρονικώς να κάνουν την υποβολή και προσπαθούμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση χάρη πλούστευσης. Βέβαια, πρέπει να κάνουμε και μια διαφοροποίηση, γιατί αλλιώς είναι 5% δημόσια επένδυση και άλλο να έχουμε 60% δημόσια επένδυση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά και μια διαφωνία με το ελεγκτικό συνέδριο. Εμεί θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ ε, μεγαλύτερου, μικρότερου ποσοστού, αλλά εν πάση περιπτώσει θα εστιαστούμε περισσότερα στα αποτελέσματα και νομίζω ότι δικαιούχος θα έπρεπε να περνά περισσότερο χρόνο να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην υλοποίηση του έργου και όχι στη χαρτούρα και στη γραφειοκρατία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ε, νομίζω ότι ένα είναι ε, σαφές για μας, για όλους μας, ότι η πολιτική συνοχή θέλει να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών και μεταξύ των κρατών μελών, βοηθά τις φτωχότερες περιφέρειες από οικονομικής, κοινωνικής απόψεως, όμως πολιτικά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ε, καταλάβουμε, αυτή είναι τουλάχιστον η άποψή μου και φαντάζομαι μπορεί και εσείς να έχετε την ίδια άποψη, η πολιτική συνοχή είναι πραγματικά το τσιμέντο που ε, συγκρατεί ε, την Ευρώπη αυτή τη στιγμή και επειδή διερχόμεθα μια τόσο δύσκολη περίοδο, πρέπει να δείξουμε ότι εργαζόμαστε για 500 εκατομμύρια πολιτών, ε, για τους δημάρχους, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, για τους πολίτες μας. Ε, δεν κάνουμε τίποτε για μας, τους αξιωματούχους των Βρυξελών. Πρόκειται για τη ζωή 500 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you. Thank you very much, Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, Επιτρόπε. Σας ευχαριστούμε για τις λεπτομερείς απαντήσεις. Πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής Κοτέρ και της Επιτροπής Ρέτζη. Και έτσι ολοκληρώνεται η κοινή συνεδρίαση στο σημείο αυτό. Πρωτού κλείσουμε όμως να δώσω το λόγο στον κύριο Όλσβα. Να κλείσει αυτό το συνεδρίαση με τα καταληκτικά του σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εν συντομία γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο που μας είχε δοθεί πάνω από μια ώρα. Εκφράσαμε πάρα πολλές ιδέες και ακούσαμε πάρα πολλές ιδέες, αλλά θα ήθελα να πω το εξή. Όλοι είμαστε φίλοι της συνοχής. Έχουμε και την ιστοσελίδα αν θέλετε να μπείτε κι εσείς σε αυτή τη συμμαχία για την συνοχή. Σας ευχαριστώ. cohesionalliance.eu Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή σας και θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα για τις περιφερειές. Ίσως θα έπρεπε όμως να συναντηθούμε και πριν από την ευκαιρία αυτή για να συζητούμε πιο τακτικά. Πρόεδρε, θα ήθελα να σας καλέσω όλους σήμερα το βράδυ, το απόγευμα, για την παρουσίαση 24 προγραμμάτων, εγώ και ο κύριος Βανίστερόι. Ξέρετε ότι είχαμε 100 προγράμματα τα οποία επιλέχθηκαν. Να σας πω ότι αυτά είναι σε όλη την Ευρώπη. Επισκέφθηκα ένα χθες. στην πλατεία. Θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρχει και μουσική. Θα βραβευτούν τα πιο δημιουργικά προγράμματα από όλη την Ευρώπη και νομίζω ότι θα είναι καλό να είμαστε όλοι μαζί για να γιορτάσουμε την πολιτική συνοχή στην πλατεία στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είναι Πολύ καλό αυτό στο τέλος της ημέρας, αλλά σήμερα τώρα θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, συμμετοχή σας και θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.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 θα πει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 Uh, Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το επόμενο σημείο της σημερινής σας διάταξης Επιτροπής ε, Ρέτζι. Πρόκειται για την παρουσίαση της μελέτης ε, που είχε παραγγείλει το Τμήμα Πολιτικής Βήτας, Βήτα για τα ε, χρηματοπιστωτικά μέσα για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια. Πριν ε, από κάποιο καιρό η Επιτροπή Έρευνα ζήτησε από το ερευνητικό τμήμα που υποστηρίζει τις εργασίες του, το τμήμα πολιτικής Β, να παραγγείλει μια μελέτη για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Όπως γνωρίζουμε, έχει προχωρήσει σταδιακά η εφαρμογή ε, το διάστημα 2014-2020. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Ευχαριστώ. Επομένως, η μελέτη έχει εξετάσει και ενδείξεις από προηγούμενες περιόδους και το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ίσχυε το 2007-2013 επέτρεπε στα χρηματοπιστωτικά μέσα να αντιμετωπίσουν μόνο τρεις θεματικούς τομείς ε, την ανάπτυξη της υπαίθρου, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενεργειακή απόδοση ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η μελέτη εξέτασε τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων για την ενεργειακή απάδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα την παρουσιάσουν οι βασικοί ερευνητές, η κυρία Φιώνα Γουίσλεϊτ, ελπίζω να προσφέρω, προφέρω σχετικά καλά το όνομά σας, και την κυρία Ρώνα Μίτσι. Είναι και οι δύο από το Ευρωπαϊκό ε, Κέντρο έρευνας πολιτικής ε, στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Έχουμε περιορισμένο χρόνο βεβαίως στη διάθεσή μας και θα ήθελα να ζητήσω να ακούσουμε πρώτα την παρουσίαση και μετά θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, δεν ξέρω ποια κυρία θα ξεκινήσει. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ Να ευχαριστήσω την κυρία Μιχαήλοβα για την εισαγωγή της και ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε εδώ για να σας κάνουμε αυτή την παρουσίαση και να σας ευχαριστήσω και για την παραγγελία της μελέτης. Ε, θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση για να παρουσιάσω τα βασικά πορίσματα και κάποιες βασικές πτυχές ε, της έκθεσης. Όσον αφορά τη δομή της παρουσίασης, πρώτα θα κάνω κάποια σύντομα σχόλια για το ιστορικό λίγο της πολιτικής και το σχετικό πλαίσιο και μετά θα σας δώσω μια εικόνα της κλίμακας της ε, στήριξης της πολιτικής συνοχής για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εν γέννη και ε, κυρίως για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Και μετά θα σας παρουσιάσω πώς ε, εφαρμόζονται τα χρηματοπιστωτικά μέσα στην πράξη. Ε, θα χρησιμοποιήσουμε και κάποιες περιπτωσιολογικές μελέτες που έχουμε χρησιμοποιήσει στην έκθεση και θα δούμε και τις προκλήσεις και τα διδάγματα τα οποία αντιλήσαμε. Και τέλος θα τελειώσω με κάποιες παρατηρήσεις για την απόδοση αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων και κάποιες συστάσεις. Το ιστορικό λοιπόν είναι σχετικά ε, σύνθετο. Έχουμε τρεις ε, σχετικές ε, θεματικές ενότητες πολιτικής. Κάθε μία είναι σχετικά περίπλοκη από μόνη της. Πρώτο, ναι, έχουμε την πρωτοβουλία Ευρώπη 2020, η οποία περιλαμβάνει στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 20% τουλάχιστον κατανάλωση και ενεργειακή αποταμίευση τουλάχιστον της τάξης του 20% για το 2030 και, ε, μάλλον συγγνώμη, για το 2030 είναι πιο φιλόδοξη ακόμα η στόχη. Το δεύτερο είναι η έμφαση στα χρηματοπιστωτικά μέσα στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν μια σειρά από πλοενεκτήματα, μπορούν να βελτιώσουν ε, την πολιτική των επενδύσεων και την ε, αποδοτικότητα ως προς το κόστος ε, των όσων δαπανούνται και έχουμε πιο βιώσιμες πολιτικές. Ωστόσο, η εφαρμογή τους μπορεί να είναι πρόκληση στην πράξη. Το τρίτο στοιχείο είναι ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Ταμείων τόσο επενδύσεων όσο και των διαρθρωτικών ταμείων. Πρόκειται για ένα νέο ε, σκέλος της πολιτικής ε, που περιλαμβάνει και τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερομένων σε ένα ήδη σύνθετο περιβάλλον. Εξετάζουμε την πολιτική για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πρέπει να γνωρίζουμε και πόσο διαφορετικό είναι το τοπίο μεταξύ των διαφόρων χωρών. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο κλίμα στην Ευρώπη που σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικές συνέπειες στην ενεργειακή κατανάλωση και στα κτίρια τα οποία είναι αυτά τα οποία κατά βάση καταναλώνουν ενέργεια. Οι φυσικοί πόροι ποικίλουν επίσης και αυτό σημαίνει ότι η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών όπως η ολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η υδροληπτική ενέργεια διαφέρουν. Ε, και επίσης ε, υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από φτωχή ενεργειακή απόδοση. Η σύνθεση ε, του πληθυσμού καθορίζει και πώς ε, μπορούμε να κάνουμε ε, εξοικονόμηση ενέργειας. Και επίσης ε, έχουμε μεγάλη ποικιλία ε, και μεταξύ αλλά και εντός των χωρών σε κάποιες περιπτώσεις. Ακριβώς λόγω αυτών των παραγόντων το τοπίο της ενεργειακής απόδοσης και την, ε, ε, ενεργεια... των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαφέρει και περιλαμβάνει και μια σειρά από πηγές χρηματοδότησης και υπηρεσίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και υποεθνικό επίπεδο. Στη σελίδα 28, αν έχετε τη μελέτη, θα δείτε ένα παράδειγμα του θεσμικού πλαισίου στη Γερμανία, το οποίο μας δίνει και μια εικόνα του πόσο σύνθετα μπορεί να γίνουν και τα πράγματα. Κάτι το οποίο είναι επίση σημαντικό είναι η κλίμακα δαπανών που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε του στόχου τη κλιματική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι είναι 100 δι ετησίω για την ενεργειακή απόδοση και 60 με 70 δι ετησίω για τι ανανεώσιμε σε επίπεδο ευρωπαϊκή Ένωση, ο πιο σημαντικό πόρος για την ενεργειακή απόδοση και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας είναι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Αν δούμε λοιπόν τώρα την κλίμακα αυτών των δαπανών λίγο πιο αναλυτικά, όπως βλέπετε από το διάγραμμα, υπάρχει ουσιαστική αύξηση στις προγραμματισμένες δαπάνες για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες στο διάστημα 2014-2020 σε σχέση με το διάστημα 2007-2013. Το 2007-2013 είχαμε 12 δις ε, στις ενεργειακές διαπάνες και ήταν περίπου το 4% της ε, πολιτικής συνοχής. Το 2014-2014 είμαστε σε πάνω από 30 δις προγραμματισμένο και είναι πάνω από το 9% της συνολικής δαπάνης. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Βλέπουμε ότι έχουμε σημαντικέ αλλαγέ μεταξύ των δύο περιόδων και όχι μόνο στι συνολικέ δαπάνε. Το 2007-2013 τα χρηματοοικονομικά μέσα τα είχαν κυρίως στόχο στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες που χρησιμοποιούνταν σε 10 χώρες. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν ε, λήφθηκαν υπόψη και πολλά προγράμματα αστικής ανάπτυξης που περιέλαμβαναν ενεργειακή απόδοση. Βεβαίω, ε, μόνο ένα μικρό ποσοστό των κονδυλίων για την ενεργειακή απόδοση και τι ανανεώσιμε ενέργειες ε, χρησιμοποιήθηκαν για τα, από τα χρηματοοικονομικά μέσα, κυρίως το 4%. Τα, η μεγαλύτερο τμήμα τη ενίσχυση ήταν μέσω επιδοτήσεων. Μέχρι το τέλος του 2015 είχαν καταβληθεί 467 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά ε, ένα μικρό ποσοστό είχε φτάσει στον τελικό δικαιούχο και στην χρηματοδότηση των έργων. Ε, δημοσιεύθηκε όμως μια συνοπτική έκθεση την προηγούμενη εβδομάδα που δείχνει ότι η απόδοση ήταν λίγο καλύτερα ε, σε επίπεδο προγράμματος από ό,τι είχε υπολογιστεί αρκετά αρχικά. Το 2014-2020 σχεδόν τριπλασιάστηκαν οι δαπάνες για την ενεργειακή απάνδοση και περίπου 20 κράτη-μέλη χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικά μέσα για τις επενδύσεις σε χαμηλή κατανάλωση άνθρακα και δίνονται 3,73 δις ευρώ και επομένω είναι ε, πολύ ουσιαστική αύξηση σε σχέση με το διάστημα 2007-2013. Είναι οκταπλάσιο. Ε, το πρώτο διάστημα όμως εφαρμογής δείχνει ότι ήταν πολύ βραδία η πρόοδος. Ε, μέχρι το τέλος του 2015 μόνο 24 εκατομμύρια είχαν φτάσει στους τελικούς δικαιούχους. Αυτό βέβαια ήταν μόνο το δεύτερο έτος εφαρμογής και μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στην επόμενη έκθεση η οποία αναμένεται εντός της χρονιάς. Βασικό χαρακτηριστικό της στήριξης για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, δείχνει ότι είναι ότι υπάρχουν πολύ ε, διαφορετικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις. Επικεντρωνόμαστε σε τέσσερις τομείς. Ενεργειακή απόδοση και στέγαση, ενεργειακή απόδοση και δημόσια κτίρια και χώροι ε, και φωτισμός δρόμων, επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες δομές και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάθε κατηγορία χαρακτηρίζεται από διαφορετικές ατέλειες στην αγορά και διαφορετική λογική παρέμβασης. Παραδείγματο χάρη, τα νοικοκυριά μπορεί να διστάζουν να επενδύσουν σε μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης, γιατί μπορεί να είναι δαπανηρά και επίσης μπορεί να υπάρχει δυσκολία ε, για χρηματοδότηση, για τα κτίρια, λόγω του κινδύνου και της πολυπλοκότητας ε, των κινδύνων. Ε, επομένως είναι τελείως διαφορετικά τα προβλήματα χρηματοδότησης για κάθε έργο σε κάθε κατηγορία. Οι λύσεις χρηματοδότησης επίσης διαφέρουν. Μπορεί να είναι η καλύτερη λύση η δανειοδότηση για επενδύσεις στο τομέα της κατοικίας και αυτό φυσικά θα μπορούσε να είναι συνήθι προϊόντα τα οποία παρέχονται από τράπεζες λιανικής, αλλά πολύ εξειδικευμένα προγράμματα κατά παρεγγελία χρειάζονται για επενδύσεις ή επενδύσεις ομολόγων σε επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα. Η μελέτη εξέτασε αρκετά παραδείγματα χρηματοπιστωτικών μέσων από την τελευταία περίοδο χρηματοδότησης. Η Εστονία και η Σλοβακία εφάρμοσαν προγράμματα ανακαίνησης ε, κτηρίων, ε, ε, ενίσχυση και εξωτερική επένδυση και μόνωση σε κτίρια και έγιναν αρκετές τέτοιες επενδύσεις και αυτά είναι για αντίστοιχης μορφής προγράμματα. Αντίθετα, στην ε, Ισπανία το πρόγραμμα Φίντες υποστήριξε τελείως διαφορετικές ε, κατηγορίες έργων. Μεταφορές, μονώσεις, εφηή δίκτυα, επενδύσεις σε δημόσια κτίρια και δημόσιους χώρους. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, εξετάσαμε μία μελέτη για ένα μέσο που επένδυε σε μικρές επιχειρήσεις που αναλάμβαναν καινοτόμα γράμματα. Και εδώ και πάλι ήταν σχετικά μικρό το ποσοστό των επενδύσεων. Πρόκειται για τελείως διαφορετικούς τύπους μέσων, λοιπόν, διαφορετικά προγράμματα και διαφορετικά όσο αριθμός των τελικών δικαιούχων. Τώρα, για την παρούσα περίοδο, έγιναν κάποιες αλλαγές ε, στους κανονισμούς που φυσικά ε, έχουν και κάποιο αντίπτυπο στις χρηματοδοτήσεις και όπως ακούσαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση πολλοί διαμαρτυρήθηκαν ότι ο κανονισμός ε, το 2007-2013 δεν ήταν ε, ε, αρκετά αναλυτικός και κατά συνέπεια είχαμε πολύ αναλυτικούς κανονισμούς για το διάστημα 2014-2020. Επικρίθηκε επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν προσέφερε αρκετές κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε έναν οδηγό με περισσότερη τεχνική συνδρομή και είχε και μια πλατφόρμα που καθόριζε και σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπήρχαν επίσης περισσότερες επιλογές εφαρμογής, ε, παραδείγματο χάρη τα μέσα ε, ε, τα οποία ήταν κομμένα και ραμμένα στα θέματα των δημοσίων συμβάσεων. Αυτές οι εξελίξεις θεωρήθηκαν από κάποιους ως βελτιώσεις μεν, αλλά υπάρχουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις. Κάποιες από αυτές τις προκλήσεις είναι αντίστοιχες ε, για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη πηγές ενέργειας ε, και σε επίπεδο επιχειρήσεων αλλά και σε επίπεδο ε, νοικοκυριών. Για παράδειγμα, το νομικό πλαίσιο θεωρείται περίπλοκο ε, οι κατευθυντήρες γραμμές καθυστέρησαν, όπως επίσης και τα πρότυπα μοντέλα, τα off-the-shelf όπως λέγονται, και γι' αυτό ακριβώς ε, είχαν και πολύ μικρό αντίκτυπο στην εφαρμογή μέχρι τούδε τουλάχιστον αυτά τα προγράμματα. Ε, τα θέματα της κρατικής ενίσχυσης επίσης ήταν δύσκολα διότι ήταν περίπλοκος ο τρόπος της χρηματοδότησης και η επιλογή των τελικών ενδιαμέσων για την εφαρμογή ε, των χρηματοπιστωτικών μέσων ήταν προβληματικός και υπήρχαν θέματα δημοσίων διαγωνισμών ε, και εμπιστοσύνης. Κάποια άλλα ήταν τα ίδια και για τα έργα χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. Εδώ είχαμε ε, συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερομένων που δεν είναι ίσως και εξοικειωμένοι με πολλούς κανόνες και συχνά υπάρχουν και τεχνικά θέματα που αφορούν τις επενδύσεις κατανάλωση χαμηλή σε άνθρακα. Και υπάρχουν κάποια τα οποία αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και ε, εξειδικευμένους ε, διαχειριστές των κονδυλίων, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο να βρούμε και ε, κάποιοι ε, διστάζουν να επενδύσουν σε αυτά, ε, προτιμούν να έχουν τελείως διαφορετική στήριξη. Όπως δείχνει και η έκθεση, το πλαίσιο, οι στόχοι και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι πολύ διαφορετικά και αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά πολιτικής από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει. Μπορούμε βέβαια να ε, αναφέρουμε κάποια ευρύτερα διδάγματα από την όλη διαδικασία. Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε και να έχουμε ένα συνολικό όραμα για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτά τα έργα ε, να δείξουμε δηλαδή τι ακριβώς γίνεται και αυτό ήταν πολύ σημαντικό σχέδιο σε κάποιες δραστηριότητες, κυρίως ε, στην Εστονία για παράδειγμα. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ευαισθητοποίηση και εδώ οι επενδύσεις ορισμένες φορές μπορεί να συμπληρώνονται και από επιδοτήσεις ε, για να γίνουν μελέτες σκοπιμότητας. Τρίτον, πιλωτικά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ε, είναι κομμένες και ραμμένες τα μέτρα τον κάθε, ε, του κάθε ε, έργου. Τέταρτον, χρειάζεται ευελιξία. Ε, πολλά από τα προγράμματα που ε, εξετάσαμε αφορούσαν αλλαγέ και μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες πολύ σημαντικά στη διάρκεια της εφαρμογή σε σχέση με τα πορίσματα που υπάρχει από την, τον προτέρων αξιολόγηση. Πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία για προσαρμογή στη στρατηγική. Χρειαζόμαστε μέτρα τα οποία θα προσαρμόζονται στις κατάλληλες τοπικές συνθήκες για να ανταποκρίνονται και στις αντίστοιχες τοπικές πραγματικότητες και τέλος, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρουμε προγράμματα από τη μια χώρα στην άλλη, είναι πολύ σημαντικό να αντλούνται διδάγματα από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους στην ίδια τη χώρα και να εξετάζουμε και τον ενεργειακό τομέα αλλά και ευρύτερα μπορούμε να δούμε ότι η εμπειρία στην εφαρμογή βελτιώνεται σύν το χρόνο. Κοιτώντα λοιπόν το θέμα τα απόδοση ε, σε ό,τι αφορά τα, τον αριθμό των προγραμμάτων για την ενεργειακή αποδοτικότητα, είναι λίγο δύσκολο να υπολογιστεί. Είναι δύσκολο να προμητρηθεί η επιτυχία οποιοδήποτε οικονομικού μέσου και επίσης είναι δύσκολο να προσμετρηθεί η υποστήριξη ε, των προγραμμάτων για ανεργική αποβατικότητα και μέσα. Άρα ο συνδυασμός των δύο είναι πιο δύσκολος ακόμα. Και ύστερα είναι σχετικά βραχυπρόθεσμη διάρκεια των ε, μέσων αυτών υποστήριξη. Ε, άρα τα αποτελέσματα θα πρέπει να τα πετυχαίνουμε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις για την καταλληλότητα των μέτρων απόδοσης, ιδιαίτερα κάποιες μελέτες αντικτύπου, ενδεχομένως να μην λαμβάνουν υπόψη κάποια από τα ωφέλη για τα προγράμματα αυτά. Για παράδειγμα, το, ε, ευρω... το σύστημα παροχή δανείων για, τέτοια, για ε, ανακαινήσεις ε, έδωσε ένα εναρκτήριο λάκτισμα, αν θέλετε, στην αγορά τη σχετική στην Εσθονία. Αυτό δεν το προσμετρούν οι τυποποιημένοι δείκτες. Η μελέτη δεν ε, περιλάμβανε συστάσεις, αλλά κάποιες προτάσεις, αν θέλετε, που προκύπτουν από την έρευνα. Και κυρίως η ιδέα ότι η προθεσμία του μέσου ενίσχυσης θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τη διάρκεια ζωής του προγράμματος. Να μην είναι τεχνητό το κλείσιμο, δηλαδή της περίοδου. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει μια περίοδος ρυθμιστικής σταθερότητας Τώρα πολλές αρχές έχουν συνηθίσει στους κανόνες αυτούς. Θα ήταν κρίμα να γίνουν ε, μεγάλες αλλαγές στην επόμενη περίοδο. Επίσης, θα πρέπει να αναπτυχθεί το δυναμικό, να ενημερωθούμε για την πολιτική και να ενημερώσουμε μέσω τεχνικής αρρωγής και σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει πιο ποιοτική αξιολόγηση των οικονομικών μέσων. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τα ζητήματα επεξεργασίας για να κατανοήσουμε τι λειτουργεί και τι λειτουργεί καλά από τα παρόντα μέσα. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την μελέτη. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα, συνάδελφοι. Έχετε το λόγο. 15 λεπτά έχουμε μόνο. Αλλά αν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο, να κάνει κάποια ερώτηση, τώρα έχετε την ευκαιρία. Everything is clear. Μάλιστα, όχι. Από ό,τι φαίνεται είναι όλα σαφή. Έχετε κάτι να προσθέσετε από την ομάδα μάλλον που κατέρχισε την έρευνα. Υπάρχουν σχόλια, προσθήκε. Um, I don't Όχι, δεν νομίζω. Ήταν ε, πολύ σύντομη αυτή η επισκόπηση που σας δώσαμε σχετικά με την ε, έρευνα. Αλλά ένα από τα στοιχεία τα οποία ανέκυψε είναι το πόσο δύσκολο είναι οι κάποιες αρχές, ε, πόσο δύσκολη είναι η χρηματοδότηση και μάλιστα πέρα από τις τεχνικές πτυχές της ενεργειακής αποφατικότητας και των ανανεώσιμων το οποίο περιπλέκει περαιτέρω τα ζητήματα αυτά για την, το σκέλο της αξιολόγησης. Ε, θα ήταν ενδιαφέρον να επισημάνουμε το εξή. Να υπάρχει μια πιο ποιοτική εκτίμηση για το πώς λειτουργούν τα εργαλεία αυτά. Δεν έχουμε σαφή ιδέα για το τι έχει αποτελέσματα και το, το τι λειτουργεί σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη ή μη των δημοσίων δαπανών. Και οι δείκτε δεν λαμβάνουν υπόψη, αν θέλετε, όλα τα φυτικά ωφέλη όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Για παράδειγμα, στο παράδειγμα τη Εσθονία, αναπτύχθηκε μία αγορά για δάνεια στον τομέα αυτό. Όπως για παράδειγμα και στην έρευνα για τους ε, ιδιοκτήτες ε, κατοικιών που θεωρούσαν ότι από την επένδυση προέκυψε αύξηση ιδιωτικού επίπεδου και ποιότητα ζωή. Αυτά δεν προσμετρούνται απαραίτητα από τους δείκτες απόδοσης. Για παράδειγμα, στο σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο μια ένα χρηματοοικονομικό μέσο το οποίο στήσονταν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για καινοτομικά προγράμματα και ένα από τα επιτεύγματα του ήταν ότι προσέλκυσε νέε επενδύσει που δεν χρηματοδοτηθήκαν απαραίτητα από τα δημόσια μέσα, αλλά τα ανέλαβε τελικά ιδιωτικό κλάδο. Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία λοιπόν, η οποία όμω δεν αποτυπώνεται απαραίτητα. Στου τυποποιημένου δείκτε απόδοση. Yeah, it was, uh, it was... Uh, ναι, λέει η Πρόεδρος. Πολύ ενδιαφέρον το σημείο αυτό και είμαι βέβαιη ότι όταν οι συνάδελφοι θα έχουν το χρόνο να εξετάσουν σε βάθος ε, την έρευνα αυτή θα ανακύψουν και άλλα ερωτήματα αναμφίβολα. Στην παρούσα φάση όμως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση, για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίασή μας. Θα συνεχίσουμε στην ημερήσια διάταξη. Που περιλαμβάνει την έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Λάμβαν παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής της ΡΕΤΣΙ της αποφάσεις των συντονιστών. εγκρίνοντα Μάλιστα. Δεν υπάρχουν σχόλια. Στα διάφορα. Η κυρία Κρέιλ ήθελε να ενημερώσω την Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις για το φάκελο Omnibus. Παρακαλώ, ενημερώστε με. Να, και εγώ κοιτώ την ομίγυρη για να δω, να μακρηγορήσω ή όχι αλλά πιστεύω ότι έχουμε και μερικούς σκιώδες εδώ μαζί μας. Εσείς είσαστε πάντα εδώ. Θα είμαι σύντομη. Προχωράμε πολύ καλά, να πούμε την αλήθεια, στους τρομερίους διαλόγους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβουλίο, το Κοινοβούλιο. Ε, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε συμβιβασμούς και αυτό μας οδηγεί σε υπερβολική ταχύτητα. Αν κατάλαβα σωστά, η budget και οι κόντα διαπραγματεύονται πολύ πιο αργά. Με πολύ πιο βραδείς ρυθμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μέσα, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, μπορούμε να πούμε ότι ναι, δεν συμφωνούμε, αλλά όλα θα πρέπει να ισουσκελιστούν και με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τον κανονισμό για τα δημοσιονομικά. Αυτό που μας ε, απασχολεί ιδιαίτερως, να τα πω κατά σειρά, είναι το ΠΑ και το, το Ταμείο Αλληλεγγύης. Εδώ δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν υπάρχει συμφωνία. Θέλαμε να απλοποιηθεί κάπως η διαδικασία. Το Συμβούλιο δεν προτίθεται να το συζητήσει αυτό μαζί μας ε, όσο δεν έχει ρυθμιστεί το δημοσιονομικό σκέλο. και αν συνεχίσουμε να παίζουμε το παιχνίδι αυτό δεν θα καταλήξουμε σε καμία συμφωνία. Γι' αυτό λοιπόν αύριο θα μιλήσω και με την κυρία Γκρέσλε η οποία είναι η αρμόδια καθήλυνα αρμόδια εισηγήτρια. Θα προσπαθήσω να το διευκρινίσω. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο, ούτε εδώ μπορούμε να πετύχουμε συμφωνία σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τα σχετικά προγράμματα. Εδώ θα ήθελα να κάνω και μια μικρή παρατήρηση. Νομίζω ότι γίνεται πολύ βαρύ λόμπινγκ από κρατημέλη, γιατί αυτό που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ότι ορίστηκε κάποιο κατόφλι ως, ε, από την Επιτροπή Ρέιτζη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι 90% όλων των προγραμμάτων ε, που βρίσκονται σε συρτάρια είναι κάτω από το όριο αυτό. Τα υπόλοιπα θα μπορούσαμε να τα ρυθμίσουμε και μετά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Επιμένω λοιπόν, επιμένω να επιμείνουμε, να εμείνουμε στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία οφείλονται σε διαφορετική μ, ρύθμιση στα κράτη-μέλη. Τι είναι δικαιούχος για παράδειγμα, πώς ρυθμίζονται τα σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά όργανα στην Ιταλία για παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι εδώ θα βρούμε συμβιβασμό, θα βρούμε συμφωνία. Και σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά μέσα, υπάρχει συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Προεδρίας, για παράδειγμα στο άρθρο 30α, όπου αναφέρεται ότι τα ταμεία ΕΖΗ χορηγούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το ΕΦΣΥ. Συμφωνούμε και θα ακολουθήσει η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, συγγνώμη, κάτι που ξέχασα να αναφέρω. Έχουμε τροπολογίες σε ό,τι αφορά τη διατύπωση με τους πρόσφυγες. Εμείς τις έχουμε καταθέσει τις ε, τροπολογίες και περίεργο πως τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Αν χρησιμοποιούσαμε την διατύπωση την οποία χρησιμοποιήσαμε στην Επιτροπή Περιφερειακή ανάπτυξη εδώ, θα μπορούσαμε... Δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε, να ενισχύουμε τα κέντρα υποδοχής των ε, προσφύγων. Αυτό δεν το επιθυμούμε ασφαλώς. Θέλουμε να μπορούμε να συνεχίσουμε να τα υποστηρίζουμε. Το επόμενο πρόβλημα που ανακύπτει είναι ότι τα ασυνόδευτα, ασυνόδευτα παιδιά, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να έχουν απαραίτητα διεθνές ε, στάτους καθεστώς, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες στα μεμονωμένα κράτη-μέλη, τις οποίες να μην τις αποκλείουμε εμείς αυτής της αρχής. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν μια διατύπωση για να τα καλύψουμε όλα αυτά. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά και με τους κοιόδες. Εγώ πρέπει να σας πω ότι κλείνω προς την αρχική διατύπωση την οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει θα διευκρινίσουμε αυτά στην συνεδρίαση με τους κοιόδες. Τώρα, υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία είναι ακόμα εκκρεμή, δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα στα δημοσιονομικά μέσα, για παράδειγμα, οι εγγύησει για απόλες τις επιδοτήσεις το θέμα της χρηματοδότησης σε προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται και από το ΕΖΕΦ και από το ESF. Είπαμε ότι η βασική ιδέα για την πολιτική συνοχή είναι να παραμείνει ένα ποσοστό τη χρηματοδότηση. Σύμφωνη η Επιτροπή, σύμφωνη και το Συμβούλιο. Θα συζητήσουμε το κατά πόσον θα το ακολουθήσουμε αυτό ω ε, γνώμονα ή μήπω θα πρέπει να βρούμε κάποιο συμβιβασμό. Ύστερα, το Κοινοβούλιο αντιλαμβάνεται ότι οφείλει να πει σε όλους τι πρέπει να κάνουν. Ψηφίσαμε μία τροπολογία εδώ στην Επιτροπή Ρέτζι, όπου ζητούμε από την Όλαφ να διεξαγάγει σχετική έρευνα. Και δηλώσαμε στην νομική υπηρεσία ότι τέτοια αρμοδιότητα εμείς ως Κοινοβούλιο δεν έχουμε. Το βγάλαμε λοιπόν. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο προκαλεί διαφωνίες και θα το συζητήσουμε ασφαλώς επισταμένως είναι το θέμα της ε, προβολής ε, των προγραμμάτων. Βλέπουμε ότι σε, όλες, σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλες τις περιφερειές δεν προωθείται, δεν προβάλλεται επαρκώς το πόσα χρήματα στις περιφερειές προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Γι' αυτό λοιπόν καταθέσαμε σχετικές τροπολογίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το, Κοινοβούλιο, και το Συμβούλιο συγγνώμη, τονίζουν ότι τους αρέσει πάρα, πάρα πολύ η ιδέα, αλλά αν θα μπορούσαμε να μην αλλάξουμε τίποτα και να μην βάλουμε και συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Να μην ε, ορίσουμε ελάχιστο προπολογισμό και ότι για παράδειγμα προγράμματα έχει ύψη και ύψου, θα πρέπει να προβάλλονται κτλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μία πρόταση την οποία, την οποία τη δέχονται πολλοί από εμά, αλλά δεν περιλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία. Αλλά θεωρώ ότι αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, και πρέπει να είμαστε σοβαροί, μια εποχή που πλήττεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από όλη αυτή την κριτική, ε, θα πρέπει να παραμείνουμε στο σημείο αυτό αμετακίνητοι. Γι' αυτό λοιπόν αυτά θα τα διαπραγματευτούμε στον τρομερή διάλογο, να δούμε πώς θα πάνε. Φαίνεται ότι θα είναι ένα πακέτο διαφιλονικούμενο. Ύστερα Σύμβουλιο και Κοινοβούλιο ε, συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή διοίκηση. Να δούμε τι θα πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικώ μήπω απλοποιηθούν τα πράγματα στο μέλλον σε ό,τι αφορά την πτυχή αυτή. Η Επιτροπή Προπολογισμού και Ελέγχου Προπολογισμών ε, θα ολοκληρώσουν, προγραμματίζουν να ολοκληρώσουν του τρεμερεί διαλόγου τον Ιανουάριο, από ό,τι άκουσα. Ε, έχουμε λοιπόν καιρό. Έχουμε καιρό και ενδεχομένω να συζητήσουμε πιο σε αρκετά ζητήματα. Γενικά, πάντως, ε, έχω να πω ότι είναι θετική η έκπληξη γιατί τα πάμε πολύ καλά και προχωράμε πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ θετικό το μήνυμά σα, γιατί είναι ένα περίπλοκο θέμα αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε τις δικές μας αποκλειστικές αρμοδιότητες και παράλληλα να διατηρήσουμε την ε, ταχύτητα και να ακολουθήσουμε την ε, κατεύθυνση που μας προτείνει η Επιτροπή Προϋπολογισμών και Ελέγχου προεπολογισμών. Αυτή είναι λοιπόν η θέση της Επιτροπής μας για τις διαπραγματεύσεις. Ε, θα συνεχίσουμε σήμερα με τη συνάντηση των σκιωδών και με τον τριμερή διάλογο σήμερα και αύριο. Αυτή ήταν η τελευταία, το τελευταίο θέμα υπό τα διάφορα. Υπάρχουν άλλα διάφορα. Ο κύριος Φανίστελρο δεν είναι εδώ. Γι' αυτό δεν έχουμε άλλα διάφορα. Να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενή μας συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 22 Νοεμβρίου του 2017 από τις 3 το απόγευμα και στις 23 Νοεμβρίου από τις 9 το πρωί. Αυτό ήταν ε, το τελευταίο πράγμα που είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς για τη δουλειά τους. Ευχαριστώ και σας. Ήταν ε, γεμάτο πρωινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα στη συνεδρία Επιτροπή Επιτροπής μας.